Θα πρέπει να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε να τροποποιήσουμε την ημερήσια διάταξη. Έχουμε προσθέσει ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη σήμερα στα διάφορα. Αφού ε, η κυρία Μαγκίνες και ο κύριος Λαβία μας είχαν ζητήσει να συζητήσουμε επί τη ουσίας ε, για τις ε, τροπολογίες της Επιτροπής μας που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προπολογισμού. Μας ζήτησαν λοιπόν να τα ξαναεξετάσουμε ελαφρώς για να τα, τις επανυποβάλλουμε στην Ολομέλεια. Εάν συμφωνείτε, να προσθέσουμε λοιπόν αυτή τη σύντομη, το σύντομη συζήτηση στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Ωραία, λοιπόν, να προχωρήσουμε με αυτήν την ε, τροποποίηση. Η σημερινή συνεδρίαση αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο. Ε, είναι επίση σημαντικό το εξή. Η συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου το απόγευμα ακυρώθηκε. Άρα παραμένει η συνεδρίαση 26 Οκτωβρίου το απόγευμα και 27 Οκτωβρίου το πρωί που θα γίνουν όπως είχε προβλεφθεί ακυρώθηκε λοιπόν το απόγευμα της 27ης Οκτωβρίου. Αυτές ε, ήταν οι ανακοινώσεις λοιπόν και περνάμε αμέσως στο workshop. Η έλλειψη πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια η λύση για ένα μακροχρόνιο πρόβλημα. Ο εισηγητής είναι ο Μάρτιν Χόσλινγκ, τον χαιρετίζω. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν είχε έλλειψη όσον αφορά τις πρώτες ύλες πλούσιες σε πρωτεΐνες για να τροφοδοτήσει τον τομέα της ε, ζωικής ε, ε, διατροφής και αυτό επιθυνώθηκε λόγω μιας ουσιαστικής μείωσης της εσωτερικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή εξαρτώμαθα ε, όλο ένα και περισσότερο από εισαγωγές. Για να στηρίξουμε την εργασία του Μάρτιν Όσλινγκ στη σύνταξη της έκθεσης για αυτό το θέμα αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτό το workshop, το εργαστήρι μέσω του Τμήματος Πολιτικής και γι' αυτό και καλωσορίζω τους συντάκτες αυτής της έρευνας, τον κύριο Ιβ Ντρόν που είναι Γάλλος και την κυρία Αλεσάνδρα Περσέ από την Ιταλία. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο και μετά από την παρουσίαση θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Παρακαλώ κύριε Ντρόν, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ε, με τιμάτε πάρα πολύ που με καλέσατε να παρουσιάσω ορισμένα στοιχεία ε, σχετικά με την εξάρτηση σε πρωτεΐνες από την Ευρώπη που είναι ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ σαν οικονομικός ερευνητής στην Ίντρα στη Γαλλία. Αυτό που θα ήθελα θα ήταν να προσεγγίσω πέντε θέματα τα οποία αναφέρονται σε αυτή την ε, έλλειψη πρωτεϊνών και να υπενθυμίσω ορισμένα θέματα σχετικά με την εξέλιξη των ε, επιφανειών και την παραγωγή των πρωτεονούχων και μετά πώς θα προστατεύσουμε τα πρωτεονούχα στις μεγάλες καλλιέργειες ε, επί επίπεδου, να δούμε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της διατροφής των ζώων στην Ευρώπη και ε, τέταρτον θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες διατάξεις οι οποίες προβλέπονται στα, πλεύμα, ε, ε, πλαίσια της εξετάσεως της κατάστασης της κοινή γεωργικής πολιτικής στην Ευρώπη και των μέτρων που ελήφθησαν στη Γαλλία για να ανακάμψουν αυτές οι παραγωγές και τέλος θα προσπαθήσω να παρουσιάσω ορισμένα στοιχεία σχετικά με το τι θα αποτελέσει ε, στοιχεία κοινοτικά που θα είναι πιο γενικά από την ε, αυτή που προβλέπετε εδώ. Στα πρώτα διαγράμματα βλέπετε την εξέλιξη των επιφανειών και ε, των ε, πρωτεονούχων καλλιεργηνών. Βλέπετε ότι μέχρι το 1993 είχαμε μία ε, αύξηση των επιφανειών, μετά είχαμε μία εξισορρόπηση μέχρι το 1998 και μετά επιμερικά μερικά χρόνια χρόνια πάλι το ίδιο επίπεδο και από το όμως το 2005 μειώθησαν σημαντικά οι επιφάνειες που έχασαν 50% εντός τριών ετών ε, βλέπετε ότι το 2009 ξανανεβαίνει η καμπύλη, δηλαδή έχουμε μία ελαφρά ανάκαμψη. Όταν λοιπόν κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες αναπροϊόν βλέπουμε ότι όλες αυτές οι παραγωγές πρέπει να αναφέρονται ε, εις ορισμένα ε, η φευρόλη είναι σημαντική και βεβαίως ε, πρέπει υπάρχει ένα βασικό θέμα ε, που τίθεται εδώ και μπορούμε να πούμε ότι ο Λουπίνος ότι η παραγωγή των πρωτεονούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιστορικά ε, ελέγχεται από τη Γαλλία που είχε τις μεγαλύτερες εκτάσεις αλλά βλέπουμε το 2009 τρεις χώρες, η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο η κάθε μία από αυτές εκπροσωπούσαν περίπου 30% της κοινοτικής παραγωγής. Εάν λοιπόν και εδώ αναφέρομαι στις 12 παλιές χώρες χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για να εξετάσουμε τις νέες χώρες βλέπουμε ότι οι τρεις χώρες που εισήλθαν το 1995 προσέθεσαν μία έκταση που τώρα αντιπροσωπεύει 70.000 ε, εκτάρια και έχουν μια σχετική ανάκαμψη ε, μετά από μια σημαντική και μετά μια σημαντική μείωση μετά το 98. Το, για τις χώρες που εισήλθαν το 2004 που έχουν μεγαλύτερες εκτάσεις 180.000 ε, εκτάρια, ιδίως με την παρουσία της Πολωνίας, αλλά και εδώ μάλλον υπάρχει μία σταθεροποίηση και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει πραγματική ανάπτυξη αυτών των επιφανειών. Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, έχουμε μία έκταση η οποία υπολογίζεται από τη ΦΑΟ στις 23.000 εκτάρια, άρα σχετικά περιορισμένη έκταση. Σε όλα αυτά τα νέα κράτη-μέλη σε σχέση με τα παλαιά έχουμε πάντοτε αποδόσεις οι οποίες είναι σχετικά χαμηλές. Συνολικά οι 12 πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εκπροσωπεύουν πάνω από το 75% των επιφανειών και το 95% παραγωγής πρωτεονούχων. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να εξηγήσουμε αυτή την εξέλιξη πρέπει να ενδιαφερθούμε για τρεις τρεις παράγοντες, η εξέλιξη της κοινοτικής ε, νομοθεσίας, ε, η εξέλιξη της αποδοτικότητος και τρίτον η εξέλιξη των τιμών. Όσον αφορά την εξέλιξη της ε, νομοθεσίας από το 72 μέχρι το 88 είχαμε ε, ε, μία ε, μία πρημοδότηση για τους χρήστες ε, ε, από το 1993 μέχρι το 2003, δηλαδή η πρώτη καμπή είναι το 1993. Δεν έχουμε πλέον μεταβλητή ενίσχυση, δεν υπάρχει κατώτατη τιμή, αλλά υπάρχει μία ενίσχυση η οποία εκφράζεται σε αξία ανατόνο και αναφέρεται σε μία απόδοση αναφοράς περιφερειακή και διαφορετική σε διάφορα προγράμματα περιφερειακής αναπτύξεως των κρατών. Όσον αφορά τα δημητριακά, υπάρχει μία μείωση της τιμής σε 9,5 ευρώ το χρόνο για το τελευταίο έτος. Από το 2004 Έχουμε μία ενίσχυση η οποία είναι πλέον σταθερή αναεκτάριο για όλες τις χώρες 55,56 ε, ευρώ αναεκτάριο και αυτή η καταποκοπή ενίσχυση ε, ε, οδηγεί σε σχέση με το παλιό σύστημα σε μειονεκτική αντιμετώπιση των χωρών και των περιφερειακών περιοχών όπου οι, ε, περιοχή, εκτάσεις αναφοράς είναι πάνω του ενός ε, εκταρίου ενώ ε, πρημοδοτούν αυτές οι οποίες έχουν χαμηλές αποδόσεις. Όσον αφορά την ανάπτυξη ε, των ε, αποδόσεων, η πρώτη, ε, το πρώτο διάγραμμα δείχνει ότι έχουμε για την Φεβρόλη μία σταθερή απόδοση, αλλά όσον αφορά τις πρωτεονούχες υπάρχει μία σταθερή μείωση και αν κοιτάξουμε τις σχετικές τιμές σε σχέση με το στάρι από πλευράς ανταγωνιστικότητος βλέπουμε ότι όσον αφορά το βάρος είμαστε στο 56% της παραγωγής του σιταριού ενώ είμαστε στο 63% της φευρόλης. Στα πλαίσια λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπάρχει ε, διαφορετική απόδοση αναλόγως των χωρών. Στη Γαλλία έχουμε έναν ε, δείκτη που είναι πάνω από το 45% σε σχέση με τον μέσο όρο της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Γερμανία είναι στο μέσο όρο, η Αγγλία ε, πιο ψηλά, ενώ η Ιταλία και η Ισπανία είναι πιο χαμηλά. Και βλέπουμε ότι εδώ και μερικά χρόνια ε, υπάρχει μία προστασία των εκτάσεων για να, ε, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχει μία οπισθοδρόμηση σε σχέση με ε, τους δείκτες του σιταριού ιδίως στις χώρες που έχουν ε, χαμηλές αποδόσεις. Αλλά μέσα σε κάθε χώρα βλέπουμε ότι υπάρχει επίσης μία μείωση του δείκτη και αυτό ισχύει για τη Γαλλία, όπου παραδείγματο χάρη έχουμε μία διαφοροποίηση 40% μεταξύ, μέχρι 40% μεταξύ περιοχών. Για να αντισταθμίσει λοιπόν κανείς αυτή τη διακύμενση θα χρειαζόταν ε, μία τιμή που να καλύπτει αυτό το 40%. Εάν δούμε λοιπόν την, ε, ε, την ε, στη Γαλλία, στη Βρετάνη βλέπουμε αφενός σημαντικές διακυμάνσεις από τη μία εσοδεία στην άλλη και ε, όσον αφορά το, ε, την τιμή και το ίδιο ισχύει και για τα είδη κουκιών και για την τιμή σε σχέση με το δίκτυ της όγιας όσο ε, αναφορά το σιτάρι έχει διακυμανθεί, διακυμανθεί χωρίς να φτάνει ποτέ το δίκτυο 1,4 που θα ήταν ε, ε, σκόπιμος για να μπορέσει κανείς να συγκρίνει την αποδοτικότητα. Δηλαδή, μεταξύ το 2006-2007 και 2007-2008 που ήταν υψηλές οι τιμές του σιταριού, είχαμε τους πιο χαμηλούς δείκτες. Δηλαδή, ε, τότε το προϊόν αυτό έγινε πολύ λιγότερο ανταγωνιστικό, πράγμα το οποίο εξηγεί γιατί η τιμή του μειώθηκε το 2008. Τι μπορούμε να πούμε ε, ότι ε, για τα, ε, τις σταθερές τιμές υπάρχει μία τιμή η οποία αντικατοπτρίζεται μέσω των ζωοτροφών και μετά προχωρά στον καταναλωτή στον ε, ε, καταναλωτή. Δηλαδή, ε, ουσιαστικά διατυπώνονται μέσω του τύπου που χρησιμοποιούν οι βιομήχανοι. Όσον αφορά το βάρος, αν κοιτάξουμε τη διακύμανσή του, βλέπουμε ότι υπάρχει μία μία σύγκριση ε, του σιταριού με τη σόγια ε, σε ε, ένα, ε, σε μια σχέση περίπου 60% πράγμα το οποίο εξηγείται από την ε, διατροφική αξία των προϊόντων αυτών όσον αφορά δηλαδή την ενέργεια. Πέραν των, ε, των σταθερών ε, των ε, διαφόρων ε, ουσιών που απευθύνονται στις ζωοτροφές βλέπουμε ότι υπάρχει μία μία ε, διαφοροποίηση μεταξύ περιοχών διότι υπάρχει η Ινδία, η Κίνα, η Αίγυπτος και μία στρέβλωση του ανταγωνισμού μέσω του Καναδά και μέ των Ηνωμένων Εθνών. Εάν λοιπόν συγκρίνει κανείς τα πρωτεονούχα σε διεθνές επίπεδο βλέπουμε ότι ουσιαστικά ε, τα πρωτεονούχα αυτά ανήκουν σε μια μεγάλη ε, οικογένεια όπου μπορούν να εναλλαχθούν και για τους ανθρώπους ε, και για την καλλιέργεια σιτηρά, ελαιούχα και ε, ε, ξηρές καλλιέργειες. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι υπάρχει μία παραγωγή 2,8 δισεκατομμυρίων τόνων που κατανέμεται ε, σε 1,2 για ανθρώπινη διατροφή και ε, το υπόλοιπο για τις ζωοτροφές. Άρα η τιμή για την ανθρώπινη διατροφή είναι πολύ σημαντική και αυξάνεται ε, όλο και περισσότερο διότι χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο φυτική πρωτεΐνη για να αντισταθμίσουμε ε, την ε, ζωική πρωτεΐνη και υπάρχει και μία δυναμική των δημογραφικών εξελίξεων και του ΑΕΠ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, το, η σόγια ε, είναι το προϊόν που χρησιμοποιείται περισσότερο, δηλαδή 280 εκατομμύρια τόνοι. Ε, αντικαθίσταται πλέον το σιτάρι από την σόγια η οποία είναι η πιο σημαντική και βλέπουμε ότι στην Νότιο Ασία ή στην Νότιο Αμερική υπάρχουν οι μεγαλύτερες εξελίξεις υπήρξε μία αύξηση της ζητήσεως των πλακών αυτών και δύο σόγια πέραν του 80% και ουσιαστικά υπάρχουν σε ε, ε, χώρες όπου ε, ε, ε, όπου η Κίνα παραδείγματος χάρη είναι πλέον ο πιο μεγάλος καταναλωτής μετά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά η Βραζιλία αλλά αυτό που έχει σημασία είναι οι εξελίξεις των και η ταχύτητά του στην Ασία όπου η κατανάλωση αυξήθηκε στο 200% σε 10 χρόνια. Στην Βραζιλία πέραν του 80% ενώ στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε σε ένα ποσοστό 1 έως 8%. Όσον, όσο δηλαδή όρημη αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, η οποία είναι μεγάλη αγορά με μικρή ανάπτυξη δεν ενδιαφέρει πλέον τόσο πολύ ε, τις εξαγωγικές αγορές ε, και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε λεπτή θέση για να μπορέσει να επιβάλλει τις τις ε, ε, δικές της ε, απόψεις από πλευράς ποιότητος όπως και για τους γενικά τροποποιημένους οργανισμούς διότι υπάρχει μεγαλύτερη πρημοδότηση από ό,τι προηγούμενα. Ε, τα πιο σημαντικά σημεία είναι, που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι αν ε, στις ΗΠΑ οι εξελίξεις είναι λιγοστές, ε, στη Βραζιλία η ανάπτυξη σταματά και δηλαδή η διεθνής αγορά βασίζεται πλέον μόνο στην Αργεντινή με όλα τα προβλήματα που μπορεί κάτι να προκαλέσει. Να σας πω κάποια τώρα στοιχεία για να πλαισιώσουμε το θέμα. Είναι περίπου 280 εκατομμύρια τόνοι με περίπου, είναι εκτιμήσεις βέβαια, έχουμε 100 εκατομμύρια τόνους για τα βοηδή ε, και 70 εκατομμύρια τόνους για τα πουλερικά και το υπόλοιπο για τα χείρους. Όλα αυτά παράγονται από τη βιομηχανία ζωικών τροφών και τα υπόλοιπα που χρειάζονται είναι υπό τη μορφή δημητριακών ή πρωτεϊνούχων ε, τροφών. Το τονάζ των ε, ε, τροφών αυτών εξελίσσεται σχετικά αργά λόγω των δύο φαινομένων, δηλαδή η βελτίωση των δικτών κατανάλωσης και από την άλλη πλευρά η πρόοδος της ε, παραγωγής ε, ζωικών τροφών, ζωοτροφών. Βέβαια τα Ε, πρόκειται για τρόφιμα τα οποία υποκαθιστούν ε, τις πρώτες ύλε με διάφορους μηχανισμούς με βάση τις τιμές και τη διαθεσιμότητα. Να σας πω και δύο λόγια για τα πρωτεϊνούχα όσον αφορά τις ζωοτροφές. Όποιο και αν είναι το τονάζ που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ποτέ, ακόμα και όταν αυτό το τονάζ είχε περάσει τους 500, τα 500 εκατομμύρια τόνους, Ποτέ δεν ε, υπήρχε πληθώρα πρωτεϊνούχων. Πάντοτε ολόκληρες οι ποσότητες απορροφώνταν και υπήρχαν και εισαγωγές που ξεπερνούσαν το 1,5 ε, εκατομμύριο τόνων. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε έναν απολογισμό για τις ε, τροφές που είναι πλούσιες σε προετίνες, οι οποίες μπορούν να υποκαθιστούν η μία την άλλη. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω εγώ αυτό τον πίνακα βεβαίως, αλλά ε, κλασικά αυτό που φαίνεται είναι ότι από την πλευρά των πόρων, από την ε, κατάργηση των αλεύρων, των ζωικών αλεύρων, η Ευρώπη εξαρτάται κατά 50% και πάνω από 50% από την κράμβη και νέα είδη ε, και από νέα είδη ηλιοτρόπιων. Έχουμε λοιπόν κράμβη κατά το μεγαλύτερο ποσοστό και οι ελαιούχοι σπόροι αποτελούν μόνο το 2%. Εάν δούμε από την άλλη πλευρά τη σόγια, έχουμε έλλειμμα στην Ευρώπη κατά 36 εκατομμύρια τόνους. Και αν μετατρέψουμε αυτά τα 36 εκατομμύρια τόνους σε επιφάνεια καλλιεργήσιμη σόγιας, αυτό σημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει περίπου 17 εκατομμύρια εκτάρια πρωτεΐνης σε μεγάλο βαθμό από χώρες της ε, Νότιας Αμερικής. Εισάγουμε δηλαδή πάρα πολλά εκτάρια για να καλύψουμε τις ανάγκες σε πρωτεΐνες. Έχουμε λοιπόν ε, τώρα έτσι μια κάποια εικόνα για το διεθνές πλαίσιο. Νομίζω πως θα ήταν σημαντικό να δούμε, αφού είδαμε την παρακμή της ε, παραγωγής πρωτεϊνών μέχρι το 2008, να δούμε αν αυτό γίνεται αντιληπτό στον έλεγχο υγείας της κοινή γερικής πολιτικής. Ο κανονισμός 73-2009 που προβλέπει ότι το πριμ για τους πρωτενούχους πόρους μπορεί να διατηρηθεί μετά από επιλογή των κρατών μελών μέχρι το 2012 στο επίπεδο του 55,57 ευρώ ανά εκτάριο όπως έχει τώρα και ότι αυτό το πριμ, αυτή η πριμοδότηση στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στο καθεστώς της ε, ενιαίας πληρωμής. Εξάλλου, υποδεικνύεται σε αυτόν τον κανονισμό ότι διατηρείται μια μέγιστη εγγυημένη επιφάνεια 1,6 εκατομμύρια εκτάρια. Είναι ιστορική επιφάνεια καλλιεργήσιμη αυτή. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν ο κανονισμός ε, ε, δημιουργεί έναν σημαντικό κίνδυνο όσον αφορά το μέλλον των πρωτεϊνούχων σπόρων, γιατί ήδη με τα 55 ευρώ ήταν δύσκολο να διατηρηθούν αυτές οι καλλιεργήσιμες επιφάνειες. Ε, άρα λοιπόν αφορσιόρι δεν υπάρχει αποσυνδεδεμένη βοήθεια, ενίσχυση. Υπάρχει το άρθρο 8 ωστόσο του κανονισμού, το οποίο αφορά την δυνατότητα ειδική στήριξης σε ορισμένες περιπτώσεις. Τρία από τα σημεία που απαριθμώνται εδώ είναι για ορισμένα είδη γεωργίας που έχουν σημασία όσον αφορά την προστασία ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Ένα δεύτερο σημείο που παρατίθεται είναι η βελτίωση της εμπορευματοποίησης γεωργικών προϊόντων και το σημείο 5 του ίδιου άρθρου λέει ότι είναι δυνατόν για ορισμένες γεωργικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν γεωργικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Και εκεί διευκρινίζεται ότι το ποσό της ενίσχυσης περιορίζεται στην κάλυψη της απώλειας ε, εισοδήματος. Και υπάρχει ένα γενικό όριο για την χρηματοδότηση στο πλαίσιο του άρθρου 68 που προβλέπεται το 10% και ένα υπό όριο για τις για εκείνες ενισχύσεις που δεν αποτελούν κομμάτι του πράσινου κουτιού. 3,5% είναι αυτό το όριο. Άρα λοιπόν η Γαλλία αποφάσισε να προστατεύσει τους ελαιούχους πόρους και αυτό το σχέδιο εντάσσεται στη συνέχεια του Γκρενέλ του περιβάλλοντος ε, και είναι ο στόχος 2020 το πρόγραμμα το συγκεκριμένο και προβλέπει ε, πέντε στόχους, έχει ορίσει πέντε στόχους, την μείωση των φυτογενομικών προϊόντων να, να, δεσμευθούν οι γεωργικές εισαγωγές μέσα στη βιώσιμη ανάπτυξη και να προσαρμοστούν οι προακτικές μέσα στην επικράτη. για τα φυτικά προϊόντα αυτό που προβλέπεται είναι η ενίσχυση της κοινοτική βοήθειας, η προστασία των ελαιούχων σπόρων μέσα στην ε, ε, ε, ανανέωση και στην ε, ε, ρύθμιση για πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την απόδοση στο στους διάφορους πόρους αλλά και αναδόμηση ή μεταρρύθμιση του τομέα των πρωτεϊνών με ανανέωση των ε, συμβατικών σχέσεων ανάμεσα στον παραγωγό και στον χρήστη. Τα μέτρα δηλαδή που ελήφθησαν το 2010 είναι μια επιπλέον ενίσχυση στους πρωτεϊνούχους ε, στις πρωτεϊνούχες παραγωγές και στα όσπρια, καθώς και βοήθεια όσον αφορά σε σπόρους αυτούς 25, ε, ανά 25 εκτάρια με την προϋπόθεση ότι, θα απομακρυνθεί αυτή η καλλιέργεια, ότι η πρώτη καλλιέργεια δεν θα αποτελεί δεν θα καλύπτει πάνω από το 45% και ούτω καθεξής υπάρχουν κάποιοι νόροι. Είναι μια ενίσχυση λοιπόν για την διαφοροποίηση των παραγωγών και αυτή η βοήθεια ε, προστίθεται στις ενισχύσεις τύπου MAE και παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά δέσμευσης για μία πενταετία. Ποιες ήταν οι συνέπειες τώρα αυτού του πρώτου σχεδίου ανάκαμψης. Ανάμεσα στο 2009 και το 2010 είδαμε μία πρόοδο 92% των επιφανειών στους ελαιούχους πόρους πάνω από 100% για τα μπιζέλια, ενώ το σύνολο των εξελίξεων των επιφανειών ήταν από το 1 μέχρι το 8%. Η γαλλική παραγωγή αυξήθηκε εν γέννη κατά 100.000 τόνους και θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε έναν υπολογισμό σε σχέση με την αποτελεσματικότητα αυτής της δέσμευσης δημοσίων κρατικών ενισχύσεων. Είναι δηλαδή 25 εκατομμύρια ευρώ που επέτρεψαν αύξηση της παραγωγής. 0,45 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή ε, κόστος 88 ευρώ το χρόνο, ε, το τόνο, συγγνώμη, όσον αφορά την ε, σόγια. Πολύ χαμηλότερο κόστος από ό,τι αυτό που αφορά το πλακούντα σόγιας. <clears throat> Αυτό αντιστοιχεί δηλαδή σε ένα κόστος περιφερειακό κατά 24% ε, κατά 24 ευρώ τον τόνο. Εάν ε, σωρεύσουμε τα κόστη, είμαστε σε ένα επίπεδο πολύ χαμηλότερο από την τιμή εισαγωγής του πλακούντα σόγια. Το 2010 επιτύχαμε το στόχο που είχε τεθεί αρχικά στη Γαλλία δηλαδή. Τώρα, σε κοινοτικό επίπεδο, το θέμα είναι να βρεθεί μια κρίσιμη μάζα ώστε να κινητοποιηθούν οι διάφοροι φορείς, είτε πρόκειται για τους ε, κατασκευαστές που παράγουν σύνθετα τρόφιμα, Δηλαδή η αγορά είναι ευρωπαϊκή με εσωτερικές ανταλλαγές που πάντοτε ήταν, ε, που ανέκαθεν ήταν σημαντικές Φαίνεται λοιπόν απαραίτητο να βρεθεί μια κρίσιμη μάζα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί ρύθμισης της αγοράς, πράγμα που δεν συμβαίνει πλέον. Ένας δεύτερος στόχος είναι η εξασφάλιση του τομέα και η ανάκαμψη της έρευνας ώστε να βρεθούν νέου, νέες ποικιλίε σπόρων και συστήματα καλλιέργειας πιο βιώσιμα και ένας τρίτος στόχος είναι να διευκολυνθεί η κάλυψη κατά των κινδύνων διακύμασης ε, των τιμών και των σπόρων. Αυτό αφορά όλες τις καλλιέργειες, αλλά είναι πολύ σημαντικός στόχος για τους πρωτεϊνούχους. Και επίσης θα πρέπει να διευκολυνθεί η διαφάνεια και οι συμβατικές ε, ε, σχέσεις μέσα στο πλαίσιο του τομέα θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ένα μέσο μία βοήθεια δηλαδή τουλάχιστον προσωρινά ανά εκτάριο για τους ελαιούχους πόρους για να αντισταθμιστεί η διαφορά ανάμεσα στο ακαθάριστο προϊόν και τα περιθώρια περιμένοντας να υπάρξουν καινοτομίες στο επίπεδο της έρευνας και της επιλογής ώστε να μπορέσει να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα των τιμών. Έπειτα αυτό που θα μπορούσαμε να προβλέψουμε είναι μία βοήθεια για την ενημέρωση για τα ωφέλη της καλλιέργειας των πρωτεϊνούχων στην προστασία του περιβάλλοντος και έτσι ώστε και οι καλλιεργητές να ενσωματώσουν περισσότερο τους υπολογισμούς για τη διάρκεια μιας ε, ε, καλλιέργειας και όχι μόνο για ένα έτος δηλαδή. Εδώ και κάποια χρόνια η βιομηχανική παραγωγή έχει απομακρυνθεί από αυτά τα προϊόντα. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο κλάδος ώστε να ενδιαφερθεί και πάλι για τα προϊόντα αυτά. Κάτι ακόμα ενδιαφέρον είναι βοήθεια να αναπτυχθούν με ε, ε, εργαλεία ώστε να προβλέπουν τις διακοιμάσεις των τιμών των ελαιούχων. Στη Γαλλία φτιάχθηκε ένα τέτοιο εργαλείο. Με συνεργασία χρηστών και παραγωγών η οποία λόγω της έλλειψης ε, μιας τέτοιας αγοράς ε, τύπου Euronex επιτρέπει να προβλέψει τις τιμές των ελαιούχων σε σχέση με την τιμή του ΣΥΤΟΥ στην αγορά αλλά μέσα θα μπορούσαν να είναι οι ενισχύσεις για την βοήθεια για τη διαφοροποίηση της αμυψης και επίσης βοήθεια όσον αφορά τις ασφαλίσεις για την σοδιά και τα εισοδήματα. Πολύ σύντομα ένα ακόμα σημείο όσον αφορά το περιβάλλον. Έχει γίνει σημαντική δουλειά στη Γαλλία μέσω της ε, του ειδικού οργανισμού για το περιβάλλον ε, όσον αφορά τα ζωτούχα λιπάσματα, την, ε, την κατάργηση της χρήσης αυτών για τις ε, διάφορες αυτές καλλιέργειες. Δηλαδή, γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την μείωση των αερίων με, που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ο κορεσμός ε, είναι πολύ μεγάλος αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα λοιπόν μία μείωση 5 τόνων στην ανεκτάριο είναι και παρόμοια η απόδοση δε στην Γαλλία. Σε σύγκριση με το 2008 έχουμε κέρδος 2,7 τόνους Ε, σε πλακούντα, πράγμα που αντιστοιχεί στο 1 εκατομμύριο εκτάρια εισαγόμενης ε, σόγιας. Επίσης υπάρχει διακύμαση των τιμών όσον αφορά τις πρώτες ύλες για τα ζώα. Διακόπτει ο Πρόεδρος στον ομιλητή, μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε με μικρότερες διακοιμάσεις τιμών Άλλο πλεονέκτημα είναι ότι τα, οι ελαιούχοι σπόροι αντιστοιχούν σε ε, συγκεκριμένες ε, χρήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την τυχητοθεσία για τα προϊόντα χωρίς ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, τα βιολογικά προϊόντα και επιτρέπουν καλύτερη αυτονομία στις πρωτεΐνες για καλύτερη γεωργική εκμετάλλευση. Τελευταίο σημείο, έχουμε κάνει έναν υπολογισμό σε σχέση με το SMG. Το οικονομικό δυναμικό των επιφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πάνω από το 2% επιφάνειας αυτών των καλλιεργιών και Επίσης, το τεχνικό δυναμικό μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι μπορούν να φτάσουν πάνω από 15 εκατομμύρια τόνους μόνο για τα σύνθετα προϊόντα. Είναι λοιπόν σημαντικές καλλιέργειες και, και ενδιαφέρουσες. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Τώρα, θα πρέπει να σας δώσω κάποια μας δώσετε σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να σκεφτούμε και τώρα ε, είναι η σειρά της κυρίας Αλεσάνδρα Πέσε του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωργικής Οικονομίας. Παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Μισό λεπτό να προετοιμάσω Okay. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τη Γενική Διευθύνση για τις ε, διαρθρωτικές πολιτικές και πολιτικές συνοχής για την πρόσκληση. Ονομάζομαι Αλεσάνδρα Πέση, εργάζομαι στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωργικής Οικονομίας που είναι ένα Ιταλικό ερευνητικό ε, κέντρο μου ανετέθη να ε, διερευνήσω πώς ε, η εξέλιξη του τομέα των πρωτενιούχων και ιδιαίτερα η εφαρμογή του mid-term review επηρέασε την ευρωπαϊκή ε, κτηνοτροφία. Δηλαδή το κομμάτι της παραγωγής με το τμήμα το τεχνικό να προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποιε είναι οι πιθανέ επιλογέ ε, από πολιτική άποψη τόσο σε αυτή τη φάση του προγραμματισμού όσο και στην αναθεώρηση 2000, μετά το 2013. Ο προηγούμενος ομιλητής μας έδωσε ένα πολύ ε, ευρύ πλαίσιο σε σχέση με τις διάφορες πτυχές ε, παραγωγής πρωτεϊνούχων την ανάλυση που εγώ έχω εκπονήσει βασίστηκα σε τρία σημεία. Δηλαδή η εξέλιξη του τομέα, η ανταγωνιστικότητα του ζωοτεχνικού τομέα και άρα και οι πολιτικές δυνατότητες, οι επιλογές. Ελέγχθη ήδη και γι' αυτό, γι αυτό το θέμα θα τα πω σύντομα, ότι υπάρχει μετά από την εφαρμογή του Midterm Review έγιναν ε, δια... σημαντικές ε, περιφερειακές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις ε, καλλιέργειες πρωτεϊνούχων προϊόντων. Υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες γνώρισαν μια πολύ μεγάλη παρακμή. Είναι οι περιφέρειες όπως ήδη αναφέρθηκε οι οποίες Ε, έχουν ε, μεγάλη απόδοση ένα εκτάριο, ενώ εκείνες οι περιοχές που έχουν χαμηλή απόδοση ένα εκτάριο έχουν μεγάλη ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα όσον αφορά τις εξελίξεις των περιφερειών, γιατί ο προηγούμενος ομιλητής αποσαφήνισε και πού οφείλονται όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις. Το πιο σημαντικό που προκύπτει από διάφορες μελέτες είναι ότι η mid-term Review του 2003 δεν τροποποίησε τις ε, επιλογές των παραγωγών. Στην πράξη, το άνοιγμα της αγοράς και άλλα, άρα ο ανταγωνισμός με άλλα προϊόντα αποτέλεσε το βασικό όχημα υποκατάστασης των παραγωγών. Σε αυτό το μικρό διάγραμμα που σας ε, δείχνω, ίσως να μην το βλέπετε καλά, προσπάθησα να αναφέρω ποιες είναι οι απόψεις των παραγωγών. Γιατί παράγουν λιγότερο Ε, πρωτεϊνούχα προϊόντα. Μέσω ερευνών που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέσω των ε, συνεντεύξεων που έχουν γίνει, σύμφωνα με το 45% των ανθρώπων που ερωτήθηκαν, η τροποποίηση έγινε μετά από το midterm review, αλλά είναι ανεξάρτητη από την τροποποίηση της mid-term review. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Αυτό το 45% ε, κάπως ε, ισοπεδώνει τις επιλογές στις διάφορες χώρες. Υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Ε, για παράδειγμα στην Γερμανία η αλλαγή των πληρωμών θεωρήθηκε πολύ σημαντική για το 54% των ερωτηθέντων. Εδώ Τώρα, σε αυτό το γράφημα, κατά κάποιο τρόπο προσπαθούμε να σας ε, κάνουμε να καταλάβετε ότι η αρχή καλλιέργειας πρωτεϊνούχων εξαρτάται καταρχήν από τα αγρονομικά πλεονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα με ψησποράς. Δεύτερον, οι τιμές ε, οι οποίες ε, ισχύουν για τις άλλες παραγωγές. Σε τρίτο βαθμό, οι τιμές που καταβάλλονται για τη βασική παραγωγή. Και τέλος, οι δύο πτυχές που λαμβάνονται υπόψη είναι η πληρωμή ένα εκτάριο και η εφαρμογή των ε, αγροπεριβαλλοντικών πληρωμών. Η μεταρρύθμιση λοιπόν του 2003 δεν στήριξε και νομίζω αυτό είναι αρκετά προφανές και από την προηγούμενη εισήγηση. Δεν στήριξε την, την παραγωγή πρωτεϊνούχων αλλά ούτε και απομάκρυνε από αυτές τις καλλιέργειες. Και κατά κάποιο τρόπο διευκόλυνε τον ανταγωνισμό όμως με άλλες καλλιέργειες. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Εάν κανεί εξετάσει τον ζωοτεχνικό τομέα και αν δηλαδή τεθεί από την πλευρά ε, των όσων χρησιμοποιούν τις πρωτενούχε ύλε για τις ζωοτροφές, Το πρώτο που προκύπτει μετά από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων που έχουμε για τον ζωοτεχνικό τομέα είναι η πολύ έντονη κρίση η οποία ταλάνισε τα τελευταία τρία χρόνια την ζωοτεχνική παραγωγή. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το περιθώριο, το μεικτό των ε, επιχειρήσεων που παράγουν ε, γαλακτοκομικά προϊόντα περιορίστηκε στο μισό από το 2007 μέχρι το 2009. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Τα τελευταία τρία χρόνια υπάρξε σημαντική αύξηση κόστους ε, όσον αφορά την ενέργεια αλλά και τις ζωοτροφές. Και φυσικά η διακύμαση των τιμών που είδαμε στην προηγούμενη παρουσίαση και στο προηγούμενα γραφήματα αποτέλεσαν τα βασικά αίτια Ο τομέας ε, ο ζωοτεχνικός ε, βαραίνει κατά 44% στην, ε, στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής, στο σύνολο της γεωργικής προστιθέμενης αξίας, το μισό δηλαδή της γεωργικής παραγωγής και η κατανάλωση ζωοτροφών το κόστος το ενδιάμεσο για την αγορά ζωοτροφών βαραίνει την αξία της παραγωγής για το 2009 κατά 54%. Η κατανάλωση ζωοτροφών 60% βασίζεται σε παραγωγή που γίνεται επιτόπου στο αγρόκτημα. 49% είναι ζωοτροφές και το υπόλοιπο είναι συγγνώμη, το 11% είναι δημητριακά που παράγονται εκεί στην, ε, στην, στο, Γεώργιο, στο αγρόκτημα και το υπόλοιπο 40% είναι σύνθετες ε, ζωοτροφές ε, που είναι όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη εισήγηση η παραγωγή η ευρωπαϊκή μάλλον παραγωγική ζωοτροφών που είχε και έχει σημαντικά ε, μερίδια της αγοράς, έχασε κάποια ανάμεσα στο 2000 και το 2008 υπέρ διαφόρων ε, αναδυόμενων χωρών όπως η Κίνα. Ας δούμε ποιες είναι οι πολιτικές επιλογές που έχουμε. Με βάση στοιχεία που έχουν προκύψει από διάφορε έρευνε, η κοινοτική πολιτική σίγουρα δεν επέτρεψε ενίσχυση του τομέα. Η ίδια η αγορά και το άνοιγμα τη αγορά μετακίνησε την παραγωγή σε περιφέρειες με χαμηλότερη απόδοση ένα εκτάριο. Το μέγα άνοιγμα στη διεθνή αγορά καθορίζει τις τιμές, ιδιαίτερα για τους τομείς εκείνους που χρησιμοποιούν τις εισαγόμενες πρώτες ύλες και κυρίως ε, στην εκτινοτροφία. Ε, έπειτα υπάρχει ένα σύστημα κάποιο, κάπως περίπλοκο, ένα σύστημα κανόνων που διέπουν τον ε, ζωοτεχνικό τομέα και που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά του. Οι πολιτικές επιλογές Ίσως να μην φαίνεται και πολύ καλά αυτό το αυτή η διαφάνεια, αλλά οι πολιτικές επιλογές που προκύπτουν από το, αυτό το πλαίσιο απορρέουν από τη μία πλευρά από τις συζητήσεις για την ΚΑΠ μετά το 2013 και ταυτόχρονα από τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις που είδαμε προηγουμένως. Τώρα, οι επιλογές για να κάνουμε κάποια διευκρίνηση επιτρέπουν να μετρήσουμε καλύτερα ποιους στόχους θέλουμε να επιτύχουμε με την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέσων ή εργαλείων η ΚΑΠ μετά το 2013 και, 13 συγγνώμη, και οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί υποδεικνύουν ότι θέλουμε να πετύχουμε διάφορους στόχους. Διατροφική ασφάλεια, ε, η επάρκεια, η διατήρηση του περιβάλλοντος, ε, η οικονομική ε, ανεξαρτησία και βιωσιμότητα, αλλά αυτοί οι στόχοι δεν συγκλίνουν πάντοτε μεταξύ τους, μπορεί να, υπάρχουν, να έρχονται και σε αντίθεση, σε αντιπαράθεση. Γι' αυτό και όταν επιλέγει κανείς την μία οδό αντί για κάποια άλλη, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η χρήση ενός μέσου μπορεί σε κάποιο βαθμό να περιορίσει την επιδίωξη κάποιου άλλου στόχου. τρεις μεγάλοι τομείς παρέμβασης. Καταρχήν, περιορισμός της διακύμησης των περιθωρίων στην εθνοτροφία που προέρχεται από τις διακοιμάσεις στις διεθνείς αγορές. Αυτό δημιουργεί, μάλλον προ, προϋποθέτει τη δημιουργία διαφόρων μέσων που θα καταφέρουν να αναχειριστούν καλύτερα το ρίσκο και που ε, θα βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των εισοδημάτων. Δηλαδή, η μεταφορά του κινδύνου μπορεί να πάει στις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές, στις ασφαλιστικές αγορές ή σε ένα πιστωτικό σύστημα που κατά κάποιο τρόπο θα το αναλάβει, θα τις αναλάβει. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά ετοιμάτων που απορρέουν από αυτή τη δομή όσον αφορά Καταρχήν, τη στιγμή όπου μεταφέρονται στην χρηματοπιστωτική αγορά με τη χρήση μέσων όπως futures, Πώς μπορεί κανείς να περιορίσει την κερδοσκοπία, δηλαδή οι τιμές να σχηματίζονται όχι από τους φορείς της αγοράς, αλλά από έμπορους, αλλά από έμπορους των futures. Καταρχήν, μια δράση μπορεί να είναι η επαλήθευση της λειτουργίας, ε, ο έλεγχος της λειτουργίας και έπειτα δεν υπάρχουν αγορές futures για όλες τις παραγωγές. ορισμένες περιπτώσεις μπορούν δηλαδή να μπουν οι προβλέψεις αυτές στην αγορά, για άλλες όχι και να υπάρχει έτσι ένας αθέμητος ανταγωνισμός για τις διάφορες παραγωγές. Η δεύτερη πτυχή αφορά την μεταφορά στον τομέα των ασφαλίσεων. Εδώ Έχουμε διάφορα παραδείγματα και ευρωπαϊκά που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το ερώτημα είναι ποιοι είναι οι άμεσοι δικαιούχοι, γιατί αν δώσουμε κίνητρα στις ασφαλίσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες ε, ε, κατά του κινδύνου. Το περίπλοκο σύστημα με το οποίο διατυπώνονται όλες αυτές οι συμβάσεις είναι ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να ελέγχεται. Για παράδειγμα στην Ισπανία το ισπανικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο ε, θεωρείται παράδειγμα γιατί το διαχειρίζεται σε μεγάλο βαθμό το κράτος. Το κράτος δηλαδή διαχειρίζεται το ασφαλιστικό σύστημα. Δεν αποκλείεται. Μπορούμε να σκεφτούμε και το καναδικό πρότυπο που είναι, ονομάζονται Agri Invest, Agri Stability, είναι δηλαδή ε, μέσα ε, χρηματοπιστωτικά όπου συμμετέχουν οι εταιρείε για να μπορέσουν να μειώσουν ή να σταθεροποιήσουν το εισόδημά τους, μάλλον, μέσω ενός πολύ ακριβού συστήματος επιχειρηματικής λογιστικής. Θα πρέπει δηλαδή να θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρότυπο οι επιχειρήσεις μας να γνωρίζουν και αυτή την πτυχή. Ένα άλλο ζήτημα όσον αφορά τα μέσα σταθεροποίησης των εισοδημάτων ή διαχείρισης του κινδύνου είναι η διαχείριση του κινδυνου μέσων ε, χρηματοπιστωτικής μηχανικής ε, και αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τη διαχείριση των επενδύσεων αλλά και για την διατήρηση των εισοδημάτων σε σταθερό επίπεδο. Στο δεύτερο πυλώνα, στην ε, πολιτική τη Γεωργική μέχρι το 2006 υπήρχε ένα συγκεκριμένο μέτρο που αφορούσε την ε, χρηματοπιστωτική ρύθμιση ή μηχανισμό ήταν ένα μέσο της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου που πλέον δεν υπάρχει, αλλά ίσως θα μπορούσαν τα ταμεία εγγυήσεων να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο. Η δεύτερη παρατήρηση είναι το να καταστεί ο τομέας της συνοτροφίας ανταγωνιστικός στη διεθνή αγορά. Υπάρχουν διάφορα μέσα, διάφοροι κανόνες, διάφορες προδιαγραφές που επιβάλλουν την χρήση συγκεκριμένων προϊόντων για την ε, τροφή των ζώων. Η ιδέα είναι λοιπόν να κατανοήσουμε πώς οι ανταγωνιστές που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές τροφικές ε, επιχειρήσεις πώς θα μπορέσουν να αντισταθούν, όπως ας πούμε διάφοροι κανόνες, όπως η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών μέσα στη σύνθεση των ε, ζωοτροφών, πράγμα το οποίο θα καθιστούσε χαμηλότερο το κόστος αγοράς της ζωοτροφής, πώς λοιπόν τα μέσα αυτά Πώς μπορεί δηλαδή η ευρωπαϊκή εκτινοτροφία να ανταγωνιστεί από τη στιγμή που υπόκειται σε τέτοιες υποχρεώσεις. βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα. Από τη στιγμή που καθορίζεται ένα σύστημα στήριξης στις ποιοτικές παραγωγές και στις ε, παραγωγές τις βιολογικές, θα μπορούσε να σταθεί ε, στον ανταγωνισμό. Και επίση, ενημέρωση σε κάθε του καταναλωτή. Χτες διάβαζα στην εφημερίδα ότι η Federal Trade Commission που είναι η πιο σημαντική ο πιο σημαντικός ελεγκτικός οργανισμός έχει αποφασίσει να συντάξει τα green guides που ενημερώνουν τους πράσινους οδηγούς, που ενημερώνουν τους καταναλωτές για όλα αυτά τα εκατομμύρια προϊόντα που υποτίθεται ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον, δηλαδή μια έντονη δυνατή στεναρή δράση για να ενημερωθεί ο καταναλωτής ώστε να έχει την στρατηγική επιλογή της ασφάλειας της διατροφικής, πράγμα το οποίο θέλει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα στοιχεία θα μπορούσαν να είναι σήματα του τύπου χωρίς ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και ούτω καθεξής. Σε πάση περιπτώσει να γίνει μια προσπάθεια ώστε οι κτηνοτροφικές ε, εταιρείες ε, και τα στάντα που πρέπει να τηρήσουν να μην αποτελούν μειονέκτημα για τον ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο. Τελευταίο στοιχείο πάνω στο οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε είναι η βελτίωση της λειτουργίας ε, της ε, ε, του κτηνοτροφικού κλάδου. Εδώ υπάρχουν διάφορα που θα μπορούσε κανείς να κάνει. Το πρώτο είναι αυτό που ήδη αναφέρθηκε, η έρευνα ώστε να υπάρξουν καινοτομίε στην παραγωγική φάση Το γεγονός ότι οι πρωτεϊνούχες παραγωγές ε, έχουν πλέον ε, θεωρηθεί ως μια ειδική παραγωγή, να μην θεωρηθούν ως να, μην πέσουμε σε ένα φαύλο κύκλο που να οδηγήσει στο ότι η έρευνα δεν ασχολείται με την παραγωγή πρωτεϊνούχων. Πάντως, όπως σας είπα, επιβάλλεται έρευνα από αυτή την άποψη. Άλλη πτυχή είναι οι συμβάσεις και η οργάνωση του κλάδου. Είναι σαφές ότι σε πολλές περιπτώσεις ότι η έλλειψη αποτελεσματικότητα στη διοργάνωση ενός κλάδου σαφώς ε, προκαλεί προβλήματα τόσο για τον παραγωγό όσο και για τον καταναλωτή. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε ποια, ποια μπορεί να είναι τα μέσα για να ε, βελτιωθεί η οργάνωση του τομέα. Στο δεύτερο πυλώνα γίνονται μελέτες όσον αφορά επενδύσεις για ολόκληρο το κτηνοτροφικό κλάδο, θα μπορούσε να είναι αυτό κάποιο εργαστήριο και έπειτα για την αναδιάρθρωση των συμβάσεων, ας πούμε οι χρόνοι, οι συνθήκες πληρωμής, οι επιπτώσεις όσον αφορά τη ρευστότητα των εταιριών, τη στιγμή που συνυπογράφουν συγκεκριμένες συμβάσεις, κάτι τέτοιο πολύ είναι πιθανό να βελτιώσει συνολικά την ε, λειτουργία του κλάδου και των επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ζητώ συγγνώμη από τους μεταφραστές αν τα πάγα γρήγορα. Ελπίζω να μην τους κούρασα πολύ. Ευχαριστώ. Tack så mycket. Eh, eh, eh, Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις τους διότι όντως τονίσατε διάφορα βασικά θέματα και βλέπω ότι πρέπει να ασχοληθούμε πολύ ε, έντονα με το θέμα των ε, λήψεων πρωτεονούχων στην Ευρώπη διότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία κατάρρευση εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις όπως παραδείγματος χάρη ε, την κατάσταση στη Γαλλία όπου επανέκαμψε η καλλιέργεια πρέπει να δούμε για ποιους λόγους τα, η, οι ε, ε, πρώτε είναι πολύ βασικές στην Ευρώπη διότι ε, η γεωργία της Ευρώπης εξαρτάται από την προμήθεια πρωτεϊνών ιδίως ε, ασχέτως του κρέατος και του γάλατος και όπως ελέγχθη υπάρχουν πολλοί νέοι παίκτες στην αγορά όπως οι Κινέζοι ε, και γι' αυτό παρεμβάλλεται και η Σόγια και εμείς δεν είμαστε πλέον τόσο σημαντικοί και γι' αυτό θα πρέπει ε, να μπορέσουμε να αυξήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την καλλιέργεια των πρωτεονούχων φυτών ε, πρέπει να ε, αναλύσουμε ακριβώς τι οδήγησε να αυξηθεί η κατάσταση αλλού Τη καλλιέργειας και αλλού να μειωθεί. Αυτό δεν μπορεί να οφείλεται στην τιμή. Πρέπει να υπάρξουν και πολιτικοί λόγοι, αν υπάρχει δηλαδή η θέληση να ε, προαχθεί. Ε, και ε, στην έκθεση την οποία εγώ καταρτίζω πρέπει να ε, δούμε ε, επίσης πώς επηρεάζουν οι διεθνείς συμφωνίες στον τομέα των πρωτεϊνών στην Ευρώπη και που πρέπει να προχωρήσουμε και των λευκομάτων διότι τα όσπρια και τα ψυχάν είναι πολύ σημαντικά και συμβάλλουν στην βιοπικιλότητα ε, διότι ε, τα, αυτά τα, ε, τα πρωτεονούχα φυτά συμβάλλουν στο να μπορέσουν να προωθήσουν την κοινή γεωργική πολιτική και να βελτιώσουν τις κλιματολογικές συνθήκες. Στην, στο συνέδριο των ΙΟΥ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 Επίτροπος τόνισε το θέμα των λευκομάτων ε, και είπε ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, δυνατότητές μας παραγωγής ε, πρωτεϊνών και πρέπει να δούμε πού μπορούμε να στηρίξουμε τη διαδικασία αυτή στο χώρο διότι ήδη αναφέρθηκε το θέμα της έρευνας, της ανάπτυξης της

Ε, και της έρευνας για νέα είδη τα οποία θα αυξήσουν ε, και ε, την προσφορά και θα ενδιαφέρουν τους γεωργούς για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε και του ανταγωνισμού των εισαγωγών. Όσον αφορά την γεωργική πολιτική η οποία διατυπώνεται μέσω αυτής της εκθέσεως έχω ήδη συναντηθεί σχεδόν με όλους τους σχεώδεις εισηγητές και νομίζω ότι δεν απέχουν οι απόψεις μας τόσο πολύ μεταξύ μας και μπορούμε να δώσουμε μία ένδειξη για μία πολιτική ώστε να καταλήξουμε σε μία συνένεση και ε, να ε, μπορέσουμε να θέσουμε σαν κοινό στόχο την, μη, την ε, κάλυψη της μειότητας των πρωτεϊνών κατά τρόπον ώστε να υποφεληθούν και οι γεωργοί και να υπάρχει μία ασφαλής γεωργία για το μέλλον για τους γεωργούς μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταμπατζή τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι η συγητής του ε, θέματος ε, για ε, την Επιτροπή Περιβάλλοντος και πιστεύω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μία απόφαση διότι σχετικά με τις εισαγωγές πρωτεϊνών εξαρτόμαστε τόσο πολύ από τις εισαγωγές ότι ώστε ή πρέπει να βελτιώσουμε την παραγωγή μας ή να αυξήσουμε την εισαγωγές κρέας κρέατο, το οποίο να απευχόμαθε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει έτσι η κατάσταση ώστε μόνο ένα τέταρτο, δηλαδή 24% περίπου των πρωτεϊνών μα, μάλλον τη καταναλώσεω πρωτεϊνών μπορεί να καλυφθεί από κοινοτικέ πηγέ, πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο διότι πρέπει να δούμε ότι η Κίνα και άλλες αγορές ε, αναπτύσσονται όλο και περισσότερο και με αυτό τον τρόπο δεν είναι πλέον δυνατόν εμείς να αυξήσουμε τις εισαγωγές μας πρωτεϊνών. Γι' αυτό και ε, με την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής πρέπει να επιζητήσουμε να ε, αποδείξουμε ότι βελτιώνεται ε, η καλλιέργεια των πρωτεονούχων φυτών παρόλο που δεν αποδίδουν όσο το σιτάρι οπότε ενδεχομένως θα έπρεπε να υπάρχουν ορισμένες ενισχύσεις όπως συμβαίνει ή στη Γαλλία διαφορετικά θα πρέπει στα πλαίσια της ανάπτυξης της υπαίθρου να προσπαθήσουμε να ε, καθορίσουμε τις τιμές κατά τέτοιο τρόπο ώστε ε, η καλλιέργεια των πρωτεονούχων φυτών να μπορέσει να έχει μία θετική επίπτωση στην προστασία του περιβάλλοντος, να μειώσει ε, ε, τα αέρια του θερμοκηπίου και να αποτελέσει μία επιπλέον πρημοδότηση για τους καλλιεργητές και τους γεωργούς. Δυστυχώς όμως αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί τώρα διότι δεν υπάρχει μία αγορά. Υπάρχει και ένα άλλο λεπτό θέμα το, τα λευκόματα της ε, ε, ζωικής προελεύσεως παρόλο που μία πρόσφατη έρευνα απέδειξε ότι ε, μπορούμε να διαθέσουμε στο εμπόριο και ε, τις φυτικές πρωτεΐνες ε, αλλά θυμάστε τι είχε γίνει στην Ευρώπη με την ε, σπογγόδη εγκεφαλοπάθεια και θέλω να αναφερθώ εδώ ή στις εισαγωγές μας των πρωτεονούχων φυτών και ζωικών πρωτεϊνών όπου 66% είναι είναι οι εισαγωγές οι οποίες είναι ε, ένα 8% μόνο της ανάγκης ε, ζωοτροφών άρα υπάρχουν ε, αναμίξεις αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των τελικών προϊόντων περιλαμβάνουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει λοιπόν κάπως να αποδεσμεύσουμε απαγορεύσουμε ε, την παραγωγή των πρωτεϊνών ε, από αυτό το σύστημα. Δεν τίθεμε υπέρ ή κατά ε, των γεννητικά τροποποιημένων οργανισμών, αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερα πρώτα πρωτεϊνούχα φυτά στην Ευρώπη. Θεωρώ την έκθεση Χόισλινγκ πολύ σημαντική. Ε, τίθεμε υπέρ αυτής της προστασίας και δεν μπορούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε ε, τα ισουσίες των εισαγωγών για, την, ε, για τις ζωοτροφές. Σας ευχαριστούμε πολύ λέει η Πρόεδρος και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Ανιώ. Sorry, Chairman. Αχ, συμπαθάτε με πρόεδρε που καθυστέρησα, γιατί είχε τεθεί ερώτηση από τον δεύτερο ομιλητή. Νομίζω ότι μπορώ να τον διαφωτίσω, να την διαφωτίσω μάλλον. Ερώτησε, τι γίνεται όσον αφορά την μη καλλιέργεια πρωτεϊνούχων, να ας πούμε για τα φασόλια, είναι το ότι τώρα έχουμε απαγορεύσει την συμμεζίνη που ήταν ένα χημικό προϊόν το οποίο σκότωνε τη χλόη που ήταν χρήσιμη και έτσι τώρα είναι εφικτό το να τα καλλιεργούμε όμως από την άλλη μεριά. Δεν θέλουν οι οργοί, ε, δεν είναι αρκετά επικερδές προϊόν, οπότε θέλουν να δουν τι γίνεται, όπως ας πούμε ε, ε, Οπότε θέλουν πιο επικερδείς ε, καλλιέργειες και πρέπει μόνο κάθε 5-6 χρόνια και επίσης κάτι άλλο σχετικά τα μπιζέλια. Είναι ότι τα μπιζέλια χρειάζονται πάρα πολλούς ε, σπόρους, πάρα πολύ ε, μεγάλη ποσότητα, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να φυδευτούν τόσο πολλοί σπόροι, ώστε αυτό είναι πάρα πολύ επιζήμιο. Το θέμα είναι επομένως το πόσο θα... Πόσο πόσο εύκολα ε, κανείς κάβει για να φυτέψει, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι και υγρό. Το έδαφος επίσης είναι το θέμα η οξύτητα του εδάφους που και αυτό είναι μια άλλη μεταβλητή. Το είδος του εδάφους επίσης όσον αφορά ε, τα, τα, τα μπιζέλια και αυτό είναι κρίσιμο. αν το έδαφος δεν είναι ε, δεν είναι μαλακό, αν έχει, πολλές, ε, αν έχει πολλές πέτρες μέσα δεν αφήνει να ριζώσει καλά. Επίσης, η ζημιά από τα περιστέρια. Αυτό έχει αυξηθεί πάρα πολύ και ακόμα και αν πει κανένα ότι ναι βέβαια Οπότε, Μάιο και Ιούνιο έχουν μεγαλύτερη μέρα, περισσότερο φως, τα περιστέρια ευνοούνται και έτσι φέρνουν πάρα πολύ μεγάλες ε, ζημιές στα μπιζέλια. Άλλο πρόβλημα. Ε, επίσης η λάσπη που υπάρχει στο έδαφος επίσης είναι πάρα πολύ ζημιογόνα. Πολλές φορές είναι κάτι άλλο το οποίο ξεχνάνε οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν αντίστοιχε κατευθυντέ γραμμέ. Νομίζω πάρα πολύ σωστά μα τα είπε ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλέ φορέ ε, οι κατευθυντήριε γραμμέ παρά είναι δημοκρατικέ και ο καθένα τι εφαρμόζει όπω τον ε, βολεύει και όπω μπορεί να προσαρμοστεί. Σα ευχαριστώ, η Πρόεδρο. Εμεί σα ευχαριστούμε. Και τώρα έχει το λόγο ο επόμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Ντοντό και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω του δύο εισηγητές για το πόσο ξεκάθαρα μα τα είπαν, ο κύριο Ντοντό και επίση να ευχαριστήσω τον εισηγητή από την Επιτροπή τη Γεωργίας. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά μαζί και όσον αφορά αυτό το θέμα με τι πρωτενε, εμεί ε, κλασικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση του να πρέπει να διαλέξουμε το πώς θα φύγουμε από, από τις παλιές συνήθειες, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις τριακόντα ετίας. θα πρέπει να δούμε πώς έχει χωριστεί η αγορά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Η Νότια Αμερική επίσης, στον πρώτο πρωτινόχα είναι μεγάλος παραγωγός και κυβέρνηση Βραζιλία και είναι σημαντικό το ότι ο βασικός πελάτης, δηλαδή η που έχουμε εμείς εδώ είναι η Κίνα που είναι πολύ πιο μπροστά από μας. Επομένως, στο μέλλον θα είμαστε μια αγορά που δεν θα ενδιαφέρει τόσο πολύ, μια που είναι τόσο απαιτητική. Δεν θα ενδιαφέρει τους παραγωγούς, γιατί αυτοί έχουν βρει μια διέξοδο πολύ πιο ανταγωνιστική για αυτούς που είναι αλλού. Αυτό θα πρέπει ομένως να μας ε, προβληματίσει, να κάτσουμε να δούμε τι γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι Όσον αφορά λοιπόν αυτές τις, αυτό, αυτό το πρωτεϊνούχα, τις πρωτεΐνες, που τα τελευταία χρονιά είναι μια, μάλλον μειοψηφία στην Ευρώπη, καλλιέργεια μειονοτική ας την πούμε, και αυτό τι πάει να πει. Πάει να πει ότι πρόκειται για μια καλλιέργεια η οποία πλέον δεν καλύπτεται από προσαρμοσμένη έρευνα για καλύτερη απόδοση. Επίσης δεν υπάρχει αντίστοιχη έρευνα τόσο ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και επίσης όπως είπε και κάποιος που έλαβε το λόγο, θα πρέπει να δούμε σήμερα πόσα χρήματα αφιερώνουμε όσον αφορά την ε, επιστημονική έρευνα για τις πρωτεΐνες στην Ευρώπη Άρα αυτά χρειαζόμαστε για να μπορεί να εξελιχθεί η παραγωγή. Είναι θέμα πολιτική ε, απόφαση που θα πρέπει να συνοδεύεται από κάποιο χρονοδιάγραμμα το οποίο να είναι ε, σταθερό και δεν μιλάω για χρονοδιάγραμμα ε, με τριετέι ορίζοντα μπορεί να είναι δεκαετή ορίζοντα και έτσι να μπορέσουμε να βρούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μας που χρειάζονται και κάποιος που λάβει το λόγο επίση, μα είπε τι έγινε στη Γαλλία πριν από δύο χρόνια θυμάμαι ότι τότε ε, είχα και μια θέση στην ε, Γεωργία και η απόφαση αυτή ξέρω ότι ελήφθη διότι οι πρωτεΐνες εμφανίζονται ως η καλύτερη λύση, η λιγότερο δαπανηρή, ούτω ώστε να καλύψουμε κάποια προβλήματα και κυρίως ε, σε σχέση με το περιβάλλον, μείωση λιπασμάτων, εντομοκτώνων και, και, και, και κυρίως θα έπρεπε κάτι να κάνουμε που δεν μπορούσε να το καταφέρουμε με τους παραδοσιακούς στόχους, στα παραδοσιακά προϊόντα. Επομένως, τώρα έχουμε μια επιλογή μπροστά μας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι πρόκειται στα μέσα επόμενα χρόνια να υπάρξει αύξηση της παραγωγής στην κεντρική Ευρώπη όσον αφορά τα σιτηρά. Και αν θέλουμε να έχουμε παραπάνω εξαγωγές δεν θα πρέπει να μείνουν σταυρωμένα τα χέρια και αλλιώς θα έχουμε αύξηση της παραγωγής. Αλλιώς θα πρέπει να σκεφτούμε μία κοινή πολιτική για το μέλλον που να φέρει μια ποικιλία στην παραγωγή και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η απόφαση για την μέλουσα ΚΑΠ να έχει και κάποια κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να βοηθά για τις πρωτεΐνες και δεν είναι θέμα διατροφής των ζώων. Είναι θέμα περιβαλλοντικό, θέμα ισορροπίας, βιοπικιλότητας που είναι πολύ ευρύτερο και σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ε, εγώ ευχαριστώ Πρόεδρε και θα πρέπει να ευχαριστήσω και αυτούς που έλαβαν τον λόγο προηγουμένως. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα και το πρώτο που έχω να σας πω είναι ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται μεταξύ σόγιας, φασολιών και μπιζελιών. Είναι κανείς όμως αν προσπαθεί τώρα να συγκρίνει πορτοκάλια με μήλα. Γιατί η σόγια για τους παραγωγούς είναι μακράν Προτιμότεροι και άρα δεν μπορούν να την υποκαταστήσουν τόσο εύκολα με τις υπόλοιπες ε, πρωτεΐνες που έχουμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα που θέλω να σας πω. Κάποιοι συνάδελφοι ανέφεραν ήδη ότι η βασική πρόκληση είναι ότι τα πρωτεϊνούχα δεν είναι τόσο ελκυστικά από οικονομικής πλευράς σε σχέση και με την παραγωγή που δίνουν άλλες καλλιέργειες. Και η τελική αποσύνδεση όσον αφορά την στήριξη, ε, μάλλον δεν θα βελτιώσει τα πράγματα. Επομένως και εγώ δεν έχω πιστεί ότι τα επιδόματα που προβλέπει το άρθρο 68 πρόκειται να θεραπεύσουν το πρόβλημα και να γεφυρώσουν το κενό και την απόσταση που υπάρχει μεταξύ θαπανών και αποδόσεων. Άρα είναι πολύ στριμωγμένη η Ευρώπη Έχουμε 35 εκατομμύρια τόνους πρωτεΐνης που εισάγουμε και η ενίσχυση στην τιμή που έχουμε είναι στο ύψος των 50 λιρών τόνο. Επομένως, υπάρχει τώρα μια έξτρα δαπάνη. 1,70 εκατομμύρια λίρες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κτηνοτρόφοι λόγω ακριβώς αυτών των προβλημάτων και της εισαγωγής της σόγιας απ' έξω. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν το έχουν οι Αμερικανοί. Εκεί δεν έχουν τους διαχωρισμούς όπως εμείς για τα μεταλλαγμένα και όχι. Η Βραζιλία είναι... έχει μεταλλαγμένα κατά 70% Στην Αργεντινή ακόμα παραπάνω όσον αφορά την παραγωγή τους. Και αυτό το κάνανε μια που είδανε τι πρεσβεύει η Κίνα και άλλοι βασικοί εισαγωγές. Δεν τους νοιάζει τι γίνεται με τα μεταλλαγμένα. Και επομένως είδαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν με την Ευρώπη ως πελάτη. Άρα έχουμε μια ορολογιακή βόμβα εδώ στην Ευρώπη. Αυτοί που μας πουλούν τα προϊόντα δεν ενδιαφέρονται. Όλο είναι και λιγότερο για την Ευρώπη. Άρα θα βρεθούμε σε συγκριτικό μειονέκτημα πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να, να εισακάγουμε ή, ή το κρέας ή το προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται για τα ζώα αυτά, το κρέας το οποίο εισάγουμε. Επομένως θα πρέπει να δούμε ότι μία από τις λύσεις είναι να αναπτύξουμε τις αντίστοιχες καλλιέργειες ή να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα και δεν νομίζω ότι το σύστημα των επιδοτήσεων βολεύει και εξυπηρετεί. Άρα ή θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις εισαγωγές, θα πρέπει τελικά τα προϊόντα στην οτροφία μας να τα εξαγάγουμε εκεί που τα ζητούν, εκεί που είναι αποδεκτά. Δεν ξέρω αν έχει το θάρρος ο Επιτρόπος Ντάλι να κάνει κάτι. Ε, είπαμε ε, δεν θέλουμε να είναι φρούριο η Ευρώπη, ούτε αυτό είναι λύση. Αυτό να στο παρελθόν και το απορρίψαμε και νομίζω θα πρέπει να μείνει σταθερή στη θέση μας εκεί, να μείνει η Ευρώπη φρούριο. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους συζητητές για την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή τους και τους συναδέλφους αλλά θέλω να περιοριστώ σε δύο σημεία. Καταρχήν την παρατήρηση ότι στη συζήτηση αυτή δεν έχει διευκρινιστεί ότι η ε, η σόγια ε, είναι ένα δευτερεύον προϊόν και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πρωτογενές προϊόν. Όπως ξέρετε η ε, σόγια αποβλέπει πρώτα στην παραγωγή ελαίου και δευτερευόντως στις ζωοτροφές και ε, επίσης οι εκτάσεις ε, αυξηθούν πάρα πολύ στο μέλλον για την ε, γεωργία διότι δεν θέλουμε μόνο να παράγουμε καύσιμα αλλά και βιοκαύσιμα και στη Γερμανία γίνεται μία προώθηση των βιοκαυσίμων δεδομένου του κόστους της γεωργίας είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει επίσης να ληφθεί η υπόψη ε, όταν εξετάζουμε τον ανταγωνισμό για την ε, ε, παραγωγή πρωτεϊνούχων. Αυτά είχα να πω προς το παρόν και προσβλέπω στην περαιτέρω συζήτηση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ντες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές, ε, τον εισηγητή μάλλον και τους ε, εμπειρογνώμονες. Πολλά έχουν ήδη λεχθεί και θα περιοριστώ σε λίγα μόνο, διότι προ τόνο είχα ε, ε, χρησιμοποιήσει ε, ζάχαρη για, δια, για ζωτροφές Γιατί, γιατί τότε υπήρχαν περισσο... μάλλον όχι ζάχαρη, μπιζέλια, διότι υπήρχε μεγαλύτερη επιδότηση και άντεχαν καλύτερα στις διακοιμάσεις του καιρού και Επίσης μπορούσαμε ε, να έχουμε ε, την ε, καλλιέργεια πολλών πολλών ε, σπόρων ε, σε ε, θερμοκήπια πράγμα το οποίο τώρα δεν υπάρχει πια. Γιατί, Γιατί λόγω της πολιτικής αποδέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως οι εγκαταστάσεις ξηράνσεως δεν λειτουργούν πλέον διότι δεν υπάρχει πλέον επιδότηση και άρα χάνουμε ε, πολλές, ε, ε, πολλές ποσότητες σπόρων που θα μπορούσαν να ξεραθούν και να χρησιμοποιηθούν ε, για τη διατροφή μας. Επίσης ε, στη γεωργία υπάρχουν διάφορες δυνατότητες ε, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της παραγωγής πρωτεονούχων φυτών αλλά αυτή τη στιγμή δεν δεν χρησιμοποιούνται και θα πρέπει να βελτιώσουμε τις μεθόδους καλλιέργειάς μας ε, των πρωτεονούχων ε, σπόρων διότι αν υπάρξει κλιματολογική αλλαγή ε, την οποία προβλέπουν πολλοί τότε θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει με κάποιο τρόπο την προμήθειά μας πρωτεϊνών και λευκομάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καπόλα Σάντους είναι ο τελευταίος στη λίστα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις εξαίρετες εισηγήσεις τους, οι οποίες επιβεβαίωσαν την δική μας εκτίμηση για το πρόβλημα. Πρόκειται για ένα στρατηγικό θεμελιώδη τομέα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία, όμως εμείς δεν μπορούμε ταυτόχρονα ενώ προσανατολίζουμε την κοινή γεωργική πολιτική στην κατεύθυνση της αγοράς, να περιμένουμε ότι οι γεωργοί θα προβαίνουν στις δικές τους επιλογές ε, για παραγωγή εκτός αυτής της λογικής και να παράγουν πρωτεϊνούχα στην Ευρώπη είναι εκτός αυτής της λογικής και γι' αυτό είμαι πολύ περίεργος ε, για τις ε, προτάσεις που ο συνάδελφος Όσλινγκ θα κάνει. Θα είναι πολύ χρήσιμες για τη συζήτηση της μεταρρύθμισης της γεωργικής πολιτικής που θα κάνουμε. Αφού δεν είναι δυνατόν να θεσπίσουμε άμεση ενίσχυση στην παραγωγή που είναι ο μοναδικός μηχανισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να προσανατολίσει την αγορά στην κατεύθυνση που εμείς θέλουμε αλλά είναι αντίθετη με τη λογική της εξέλιξης της ΚΑΠ και των ε, αποφάσεων που λάβαμε με τις έκθεση του συναδέλφου Λάιον άρα η μόνη δυνατότητα για να διατηρηθεί κάποιο κίνητρο είναι μέσω ενός μέτρου τύπου ε, του άρθρου 68. Ειλικρινά, εγώ δεν έχω φαντασία για να προχωρήσω περισσότερο και δεν είδα μέχρι τώρα και καμία εναλλακτική ε, ε, πρόταση πιο εφάνταστη και γι' αυτό και πραγματικά Περιμένω πολλά από το συνάδελφο, να δούμε αν δεν έχει δηλαδή αρκετά ζωηρή φαντασία για να προβλέψει κάποιο μέτρο το οποίο να αντιστοιχεί στις δικές μας προσδοκίες αλλά και στην κατεύθυνση που ακολουθεί η κοινή γεωργική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, οπότε με αυτή την παρέμβαση ολοκληρώνεται η συζήτησή μας, για να δεν κάνω λάθος. Α, όχι. Όχι, όχι, όχι. Συμπαθάτε με. Βεβαίως. Θα πρέπει να λάβουν το λόγο ξανά οι εμπειρογνώμονες και να απαντήσουν τις τεχνολογίες που τους υπευλήθησαν. Έχετε το λόγο. Ναι, όντω θα πρέπει να γίνουν ε, κάποιε διευκρινήσει σε σχέση με τα θέματα τη ενισχύση στα προϊόντα το, το και βεβαίω και το θέμα δεν υπάρχει πάγια βοήθεια. Αλλά θα πρέπει να καλύψουμε τον κίνδυνο για την επόμενη διετία ή τριετία. Δηλαδή και κατά πόσον ε, απειλείται με εξαφάνιση η παραγωγή. Είναι σημαντικός ο κίνδυνος ότι δεν είναι δυνατόν μετά να επανέλθει στα προηγούμενα κατάσταση. Επομένω, χρειάζονται κάποια μέτρα εν αναμονή των ε, αποτελεσμάτων της ε, έρευνας για τους νέους σπόρους. Υπάρχουν μεγάλα προγράμματα που αφορούν αυτά τα προϊόντα και θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση γιατί το διηγήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τα όσπρια Ινδία, Πακιστάν, Αίγυπτος, το διεκείμενο είναι ευρύτερο από την Ευρώπη. Εκεί είναι πολύ σημαντική τροφή. Άρα σε διεθνές επίπεδο γίνεται ιδιωτική έρευνα η οποία δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ πέρα από τον Καναδά. Οπότε Γι' αυτό ακριβώς και η Ευρώπη μπορεί να δραματίσει σημαντικό ρόλο μια που είναι όλες αυτές οι μεγάλες χώρες, είναι παραγωγή οσπρίων και έχουν ελληματική παραγωγή. Μια που η εγχώρια παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει ε, την ζήτηση από τον πληθυσμό. Επομένως από αυτή τη πλευρά μπορεί να διαπτύσσει κάποιο ρόλο η Ευρώπη εάν είναι αυτάρκης όσον αφορά την παραγωγή της και έτσι ίσως είναι δυνατόν να καλύψει το προσωρινό έλλειμμα και να έχει έτσι και μεταφορά καινοτομία και τεχνολογία. Ringrazio innanzitutto tutte le persone che sono intervenute e le sollecitazioni. Να ευχαριστήσω όλου που παρενέβησαν και για τα όσα είπαν, για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε σε κάποιε από ε, σε κάποια θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την Κομισιόν. Εγώ ανέφερα τρία κεντρικά ζητήματα. Καταρχήν, έχουν γίνει πολλές, κάποιος με, ρώτησε πόσες έρευνες έχουν γίνει για τις ελαιούχους πόρους. Δεν θα ήταν άσχημο μάλιστα να γίνει μια επαλήθευση για το τι ακριβώς είναι έρευνα, ορίζεται ω έρευνα σε αυτό το τομέα. Επίση θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ωστόσο ότι πολύ συχνά η έρευνα εγκαταλείπει, όπως είπε και ο συνάδελφο τα θέματα και τα επιχειρήματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο μπορεί να αφορούν μόνο μια μικρή παραγωγή ή μια πολύ συγκεκριμένη δικευμένη παραγωγή. Δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος. Ίσως λοιπόν η Κομισιόν θα μπορούσε να κατευθύνει τις ερευνητικές ε, δραστηριότητες προς την κατεύθυνση αυτών των ε, προϊόντων. Έγινε λόγος για την παραγωγή των βιολογικών καυσίμων ε, από μια έρευνα που έγινε το 2009 είναι προφανές ότι η υποκατάσταση αυτών των παραγωγών από τα βιολογικά καύσιμα είναι άμεση, είναι προφανής. Σταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ορισμένα προϊόντα που έχουν ε, στόχο την ενέργεια, την παραγωγή ενέργειας μπορεί στην υποπαραγωγή τους να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές. Άρα λοιπόν Κατά συνέπεια, η καθαρή επίπτωση είναι ναι, υποκατάσταση των πρωτενούχων, αλλά ταυτόχρονα η χρήση ορισμένων υποπροϊόντων της παραγωγής ε, των, ε, των, των ενεργικών παραγωγών που μπορεί κατά κάποιο τρόπο να διευκολύνει την ε, εσωτερική παραγωγή όσον αφορά την χρήση για τις ζωοτροφές. Αφορά Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο του είδους αυτού της παραγωγής ότι πρέπει να υπάρχει ανεχνεσιμότητα του προϊόντος. Είναι προφανές ότι από την άποψη της ασφάλειας του προϊόντος και της ενημέρωσης του καταναλωτή Αυτό αποτελεί ένα μέτρο πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όσον αφορά τις βιολογικές παραγωγές. Πολύ πιθανόν είναι ότι μια δράση σε αυτό το, από αυτή την άποψη θα μπορούσε να προσανατολίσει την ίδια τη βιολογική παραγωγή. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και τους δύο εμπειρογνώμονες γιατί να σας δώσω μια πάρα πολύ καλή εικόνα του τοπίου και το να δώσουμε τον λόγο στον εισηγητή, αν θέλει βεβαίω να υποβάλει κάποιε παρατηρήσει σε σχέση με αυτά που ακούσαμε από συναδέλφου και προγνώμε. Κύριε Χόστιν, έχετε το λόγο. Ναι, θα παρουσιάσω την έκθεση στην επόμενη συνεδρίαση. Βέβαια ε, θα ενσωματώσω όλες τις προτάσεις και υπάρχει ένα πράγμα που με κάνει πιο επιφυλακτικό ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ε, καταρχήν το πρόβλημα είναι αμφιλεγόμενο και είναι ε, ένα σημείο κινήσεως στην πολιτική για να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση. Επίσης ελέγχθη ότι θα πρέπει πρέπει στην γεωργική πολιτική να ληφθεί υπόψη και το θέμα αυτό. Δεν θέλουμε δηλαδή να δημιουργηθεί μία νέα προνομιούχα θέση ε, ε, στη γεωργική πολιτική αλλά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο αυτό στο μέλλον για να αποτελέσει βασικό σημείο της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής η οικονομική πτυχή θα πρέπει να συνδυαστεί ε, εις ε, ε, τον τομέα των κρεατοπαραγωγών και με την μεγάλη οικολογική χρησιμότητα αυτής της φυτικής παραγωγής πρωτεϊνούχων διότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει όλοι να συμβάλλουμε. Ε, είμαι όμως επιφυλεκτικός προς το παρόν. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τους χιώδεις εισηγητές κατά τρόπον ώστε ε, να βρούμε μία κοινώ αποδεκτή λύση με πολλή φαντασία, ενέργεια και προσβλέποντας ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Δεν ξέρω τώρα μήπως πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο, δηλαδή στην παρουσίαση πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, έχουμε τον εκπρόσωπο εδώ τη Επιτροπή. ναι. Είχαμε προγραμματίσει να αρχίσουμε στις 5 η ώρα. Ε, μιλούμε για την ηλεκτρονική αναγνώριση των προβάτων. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και είναι καυτό για πολλά μέρη στην Ευρώπη. Επομένω, να δώσουμε ευθύ αμέσω το λόγο στον εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν είναι εδώ. Ο εκπρόσωπο ή εκπρόσωπο δεν ξέρω. Έχετε το λόγο πάντω. Come i membri del Parlamento sicuramente ricorderanno. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Όπω ε, σίγουρα θα θυμούνται οι Ευρωβουλευτέ, ε, κατά τη διάρκεια του 2003 και 2004 υιοθετήθηκε μια νομοθεσία σε σχέση με το νέο σύστημα εντοπισμού και αναχνευσιμότητα των, των προβάτων. Αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας τρομερής κρίσης, εκείνης της κρίσης ε, της επιζωτίας του αυτόδου πυρετού που χτύπησε σε διάφορα κράτη όσον αφορά την εκτινοτροφία και τα συγκεκριμένα είδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έφτιαξε ένα σταδιακό σύστημα εφαρμογής των νέων κανόνων. Σε αυτή τη φάση, από την 1η Ιανουαρίου 2010, ενεργοποιήθηκε το σύστημα και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία. Βρισκόμαστε ωστόσο ακόμα σε μια σταδιακή φάση εισαγωγής του συστήματος. Το σύστημα εντοπισμού και ανιχνευσιμότητα ε, μεμονωμένη των προβάτων θα πρέπει να ε, τεθεί τελικά πλήρω σε λειτουργία από την 1η Πρώτη 2012. Έχουμε λοιπόν ακόμα 15 μήνε μπροστά μα για να, πώς να το πω, τελειοποιήσουμε το σύστημα η Κομισιόν ευνόησε μια σταδιακή εφαρμογή του συστήματος με μια ολόκληρη σειρά μέτρων ε, γνωρίζοντας ακριβώς πως αυτό το νέο σύστημα θα ήταν ε, ιδιαίτερα βαρύ για εκείνα τα κράτη-μέλη που εκτρέφονται πολλά εγωπρόβατα. Αυτή τη στιγμή ελέγχουμε την εξέλιξη της κατάστασης. Έχουμε συζητήσει με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στο πλαίσιο της μόνιμης Επιτροπής για την Διατροφική Ασφάλεια και την Υγεία των Ζώων και προέκυψε ένα πλαίσιο το οποίο θα προσπαθήσω να σας ε, παρουσιάσω συνοπτικά. Καταρχήν, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται για την εφαρμογή του συστήματος και τα περισσότερα κρατημέλη είπαν ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει ιδιαίτερα τεχνικά προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος. Θα πρέπει μάλιστα να πω ότι ακόμα και όταν το σύστημα εντοπισμού των βοηδών ξεκίνησε, Υπήρξαν κάποια προβλήματα, αλλά πιστεύουμε πως ε, και τώρα θα ξεπεραστούν μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Φυσικά υπάρχει ακόμα μια αντίσταση από πλευράς ορισμένων ε, κτηνοτρόφων που σχετίζεται και με το κόστος του μικροτσίπ. Το κόστος ε, των διαφόρων σημάτων των ηλεκτρονικών. Ε, ειδικά συστήματα είναι αυτά που τοποθετούνται στα αυτιά των ζώων, αλλά ε, στα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν πολλά εγωπρόβατα και όπου οι παραγωγοί κατάφεραν να αποσπάσουν καλύτερες τιμές σε σχέση με τα μικρότερα κράτη-μέλη όπου ο αριθμός των εγωπροβάτων είναι μικρότερος. Ορισμένα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν δημόσιο χρήμα για να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους στην εφαρμογή του συστήματος. Μα μόνο ένας περιορισμένος αριθμός χρησιμοποιεί το κονδύλια της ανάπτυξης του Ισυπέθρου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των κοινωτικών ε, χρηματοδοτήσεων. Αυτό σημαίνει πως ορισμένα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν κυβερνητικά κονδύλια, κρατικά κονδύλια. Για την ώρα τα κράτη-μέλη δεν μας έχουν υποδείξει προβλήματα σε σχέση με τις κυρώσεις ε, για την ε, συμμόρφωση. Υπάρχουν ομοιόμορφες ε, Ε, διατάξεις και υπάρχουν ε, προβλέψεις για κυρώσεις Ωστόσο, ακόμα δεν μπορούν να επιβληθούν λόγω του ότι το σύστημα δεν έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Η Κομισιόν προσέχει ιδιαίτερα το θέμα και γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον σε ένα κράτο μέλο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν πολύ έντονε αντιστάσει. Κατά τη γνώμη μου αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο ε, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο μετακινούνται τα εγωπρόβατα πολύ συχνά σε ε, τμήματα που αποτελούνται από μικρά ζώα από το ένα αγρόκτημα στο άλλο και η... χρησιμοποιείται η αγορά γιατί εκεί τα ζώα αναμειγνύονται, δημιουργούνται νέες ομάδες ζώων που έχουν διαφορετική προέλευση και μετά Αυτά τα ζώα, αυτές οι ομάδες στέλνονται στις ε, διάφορες ε, στα αγροκτήματα. Σε ένα τέτοιο σύστημα, οποιοδήποτε εφαρμογή ενό σοβαρού προγράμματο ανεχνευσιμότητας θα είχε να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Την επόμενη εβδομάδα οι εμπειρογνώμονες της Κομισιόν από την Γενική Διεύθυνση Υγεία και Καταναλωτές όσο και από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας θα μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να δουν από κοντά αυτού του είδους τα προβλήματα και να διερευνήσουν τι είδους ενέργειες θα μπορούσαν να κάνουν και μια ανησυχία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η πολλαπλή συμμόρφωση. Και ως προς αυτό είπα πριν από τρεις μήνες σε αυτή την Επιτροπή ότι σε σχέση με τον εντοπισμό των ε, βοηδών, η Κομισιόν, επαναλαμβάνω, όσον αφορά τον εντοπισμό των βοηδών, η Κομισιόν έχει ήδη δεχτεί την αρχή πως η κτηνοτρόφοι δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν για τις ελλείψεις ε, ή τα μειονεκτήματα του ίδιου του συστήματος και όχι δικές τους παραλήψεις ε, ή έλλειψη βούλησης εφαρμογής του συστήματος. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εφαρμοστεί αυτή η αρχή και σε σχέση με τον εντοπισμό, ε, τον εντοπισμό και την ανεχνευσιμότητα των εγωπροβάτων. Επαναλαμβάνω ότι έχει προβλεφθεί αποστολή από την DJ Sanko και την DG Επιπλέον, το, η υπηρεσία ε, τροφών και κτηνιατρικής έχει προβλέψει αποστολές σε διάφορα μέσα στη διάρκεια του 2011 ακριβώ για να προβεί στην επαλήθευση της λειτουργίας του συστήματος και είναι σαφές ότι επί τη βάση των πληροφοριών των πρόσθετων που θα έχει θα μπορέσει η Κομισιόν να φτιάξει εκείνα τα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να εγγυηθούν με τη σειρά τους στη σωστή εφαρμογή του νέου συστήματος εντοπισμού και ανιχνευσιμότητα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα ευχαριστούμε κύριε Λαπομάντα και ξεκινάμε τη συζήτηση. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Ο Τζέιμς Νίκολσον έχει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν περίμενα να είμαι ο πρώτος που θα δώσετε το λόγο. Πάντως άκουσα με τεράστιο ενδιαφέρον τον ε, ε, κύριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος μας τα είπε και δεν ξέρω ακριβώς πού πληροφορηθήκατε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τουλάχιστον στη μετάφραση αυτό πέρασε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, άκουσα επιλέξει. Και είπατε ότι υπάρχει κάποιο αντίσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να Σήμερα το πρωί ήρθα από την περιφερειά μου τη Βόρεια Ιρλανδία και τι να σας πω. Υπάρχει πρόβλημα για την εφαρμογή αυτής της ε, ηλεκτρονικής αναγνώρισης. Και το πρόβλημα είναι ότι η τεχνολογία δεν έχει ακόμα τα στάνταρ που χρειάζονται ούτως ώστε να αποδώσει. Πώς, πώς θα το κάνω αυτό επί τόπου. Πολύ ωραία μπορεί να κανείς να το πάει στο, στο, σχετικό τόπο το ζώο και οπότε εκεί πέρα μπορεί να ε, ε επισημαθεί, μπορεί να, να το μαρκάρουν. Αλλά όμως μετά στην επόμενη ε, φάση τα χάνεται το σημάδι και έτσι δεν έχουν ταυτότητα τα ζώα και δεν φταίει το ζώο. Η τεχνολογία αυτή που δεν επαρκεί. Και τώρα φτάνουμε στην κατάσταση κατά την οποία οι κτηνοτρόφοι έχουν ξοδέψει ένα σωρό λεφτά για να μπορούν να έχουν το σύστημα της αναγνώρισης και της ανάγνωσης αυτών των ετικετών ας πούμε και ξέρετε δεν ζήτησαμε εμείς να ζητηθεί το θέμα σήμερα το ζήτησαν άλλοι συνάδελφοι και ξέρετε γιατί, γιατί εγώ θεωρώ ότι η μάχη χάθηκε. Είναι τόσο ηλίθιο το σύστημα που είναι ανεφάρμοστο. Κάθισα και μίλησα με τον κόσμο. Ιδίω με εκείνου που έχουν καλή ράτσα ζώα, πρόβατα και μου είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα καλό μεταχείριση των ζώων γιατί μετά από κάποια χρόνια δημιουργείται μόλυνση στα αυτιά των ζώων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πονάει το ζώο. Ενώ το άλλο σύστημα όπου οι κτηνοτρόφοι βάζανε κάποιες απλές πλαστικές ετικέτες δεν έφερνε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Τους πρίζεται το αυτοί, υποφέρουν τα ζώα. Ε, γιατί λοιπόν να κάθονται να υποφέρουν τα ζώα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι τρομερό από πλευρά καλών των ζώων. Ωραία, έγινε ό,τι έγινε. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και θα ήθελα στα σοβαρά να δούμε τι γίνεται επί Και να δείτε και εσείς πληροφορίες που παίρνετε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπά και σας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ε, τότε αυτό σημαίνει δεν έχουν ιδέα με το τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στο κράτος τους. Άρα, πηγαίνετε επί τόπου, μιλήστε σε αυτούς που εφαρμόζουν το σύστημα, και καμιά φορά ξέρετε δεν το πολυδάπανο είναι το να πάει κανείς πίσω αντί για μπροστά. Γιατί θυμάμαι σωρό κόσμο πριν από τρία-τέσσερα χρόνια είχε αντεπιχείρημα για αυτό το σύστημα. Εμεί τα λέγαμε, οι άλλοι λέγανε ότι δεν πειράζει. Να τώρα έρθει η ώρα τη εφαρμογή και τώρα κατάλαβε ο κόσμο πόσο δύσκολο είναι αυτό να υλοποιηθεί. Ακριβώ διότι τα, τα, τα εγωπρόβατα συνήθω είναι σε κάποιε περιοχέ ε, ε, που είναι, σε, είναι, είναι ε, είναι ορεινές περιοχές, είναι, ε, είναι, είναι, είναι πάνε εδώ στους, στους, στα φαράγγια, στα λιβάρια, που, σε, διάφορα ε, κρύβονται από εδώ, από εκεί, τι να σας πω, πού να τα μεταφράσουν για αυτά οι δημιουργίες, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει, ε, όσο θα πρέπει να σας πω, να καταλάβετε ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα σημειωθεί κάποια πρόοδος, δεν ξέρω, και ε, θα έρθουν και θα μου πούν εμένα Ήδη κτηνοτρόφοι. Τι έγινε, γιατί ξέρουν τόσα λεφτά αφού έχουμε τεχνολογία ε, που, που, που δεν μας βοηθάει. Οπότε, εάν δεν ε, κάνουμε αυτό που πρέπει στην τεχνολογία αυτή που δέχεται βελτιώσει, δεν κάνουμε τίποτε. Καλά. James, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αντιπρόεδρος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε και εμένα ήρθε και με βρήκε κόσμος από κάτω χώρες, Βέλγιο, Γερμανία και μου είπαν παρόμοια αυτά που είπαν και στον Τζιμ τα προβλήματα αυτά τα οποία αντιμετωπίστηκαν και στον Βασίλειο σε σχέση με το κόστος, σε σχέση με την γραφειοκρατία, σε σχέση με το ότι πρόκειται για σπατάλη χρόνων. Και ήρθε ένας Ολλανδός στο γραφείο μου κάθε στο γραφείο μου, άνοιξε τον υπολογιστή μου και μου έδειξε τι βήματα πρέπει να κάνει ώστε να μπορέσει να μπει στο σύστημα για να ε, το εφαρμόσει. Το σύστημα όμως δεν λειτουργεί, επομένως ο κόσμος έχει πρόβλημα. Δηλαδή, τελειώνει τη δουλειά του στο χωράφι, γυρίζει σπίτι γιατί να ξεκουραστεί που ξεκουράζεται, α πούμε, ο σκύλο του που τον συνοδεύει. Πρέπει να κάτσει στον υπολογιστή πάρα πολλή ώρα για να μπορέσει να εφαρμόσει το σύστημα αυτό. Δεν ξέρω τι είχαν πει οι Κομισιόν, αν μπορούμε να το βεβαιώσει. Το σύστημα όμω είναι ατελέ και θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο καλύτερα θα μπορούν να μπουν τα δεδομένα στο σύστημα, πώ θα εισαχθούν. Γιατί αν θέλει να, να, να, να, να μπει σε μια τράπεζα δεδομένων και να πάρει κάποια δεδομένα ο κάποιο ε, κτηνοτρόφο όσον αφορά το, τον τόπο που βρίσκονται τα πρόβατά του, ε, κάπου παραπέρα, τέλο πάντων, άμα έχει περάσει τα, τα σύνορα, α πούμε, ο συγκεκριμένο έξω από την Ολλανδία, δεν μπορεί να πάρει αυτέ τι πληροφορίε. Το σύστημα τον αφήνει να, να, να πάρει δεδομένα εκτό ορίων ε, χώρα. Επομένω, αυτά ήρθαν και μου είπαν. Ε, η κατάσταση είναι δραματική και ε, συμφωνώ με τα όσο είπε ο κύριος Νίκολσον ότι εμείς καθόμαστε εδώ και τα κουβεντιάζουμε, όμως οι κτηνοτρόφοι είναι πάρα πολύ θυμωμένοι και δεν νομίζω ότι το πρόβλημα τελικά είναι πρόβλημα που υπάρχει μόνο στο Ηνωμένο ε, Βασίλειο. Είναι πολύ ευρύτερο γιατί έχω ακούσει παράπονα και από άλλα τρία κρατημέλη και για αυτό έχω κάτσει και έχω συντάξει κάποιο είδου διαδήματα ε, και με χαρά μου βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξετάζει, το μελετά και ότι η, Ευρω... Επιτροπή μας επίσης το συζητεί μια που το πρόβλημα είναι υπαρκτό και προβληματίζει τους κτηνοτρόφους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιπρόεδρε. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ανιώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ περίπλοκο είναι το θέμα. Πάρα πολύ πολύπλοκο να το συζητήσεις, ακόμη πιο πολύπλοκο για να το, να το διαχειριστείς επί τόπου. Σε αρχή της ξεκίνησε το θέμα και το θέμα ήταν τι θα γίνει με τα αρνιά εκείνα τα οποία μεγάλωναν σε μία εκμετάλλευση και μετά έπρεπε να πουληθούν σε κάποια άλλη εκμετάλλευση γιατί εκεί πέρα υπήρχε κατάλληλη κατάσταση για να βγάλει το χειμώνα, το χυμαδιό ας πούμε. Ε, Επίση, ακριβώ το πρόβλημα ήταν ακριβώ για, για τα αρνιά τα οποία πρέπει να μετακινηθούν από λοφόδες ή μειωρινέ περιοχέ ε, σε κοπάδια των 20 και κατόπιν θα έπρεπε να, να, να, να, να μπουν σε κάποιες φραγμένες περιοχές για να τα εξετάσουν οι, οι αγοραστές και μετά πρέπει να γυρίσουν πίσω στο Μαντρί. Στο Άσφορντ έχουμε 8.000 τέτοια αρνιά, τα οποία μέσα σε μια μέρα πρέπει να σε αυτή τη διαδικασία και μπορεί να πουλήσει 20 τέτοιες περιοχέ περιοχές, διαφορετική την διαθεμία ο κάθε Τώρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με κάποιες ομάδες ε, θηλυκών ε, αμνών που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή. Είναι πάρα πολύ ακριβά, χωρίζονται, πουλούνται χωριστά από τους εκδημοτρόφου γιατί ε, κάποιοι θα αγοράσουν μόνο τέτοια και θα πρέπει να υπάρχει ένα, μια ετικέτα και να μπορεί να τη διαβάσει ε, κανείς ηλεκτρονικά το, οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί τα, τα πρόβατα πάνε πέρα δόθεμε στην περιοχή μερικά ε, χαμηλώνουν το κεφάλι τους, μερικά το βάζουν κάτω από ένα άλλο αρνί και πολλές φορές λοιπόν είναι δύσκολο να γίνει ταυτοποίηση, πολλές φορές πηδάνε, πολλές φορές ξεφεύγουν ε, τρυπώνουν από εδώ από εκεί, πηδάνε πάνω από το, από το φράχτη και άντε να τα βρεις τώρα μέσα στην αγορά που γίνεται χαμός. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα δοθεί χωριστό χρώμα ε, σε κάθε πρόβατο που είναι σε συγκεκριμένο φράχτη, μικρό μαντρί στην αγορά που είναι διαφορετικό από τα άλλα μαντρία στην περιοχή και οπότε κάθε φορά έχουμε τέσσερις ε, εργάτες οι οποίοι πρέπει να κάνουν αυτή τη ε, δουλειά. Όμως η δουλειά δεν μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε. Θα πρέπει να είναι αυτοί πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Αυτό πάει να πει ότι έχουν ψηλές δαπάνες, μετακυλίονται στην τιμή του αρνιού και επομένως ε, έχουμε τώρα διπλάσια γραφειοκρατία από ό,τι πριν μου είπαν οι κτηνοτρόφοι ότι θα πρέπει να έχουν όλα αυτά τα χαρτιά όταν κάνουν τις, δουλειέ τις, τις δουλειές αυτές. Ε, ένα σωρό αρνιά χάνουν τις ετικέτες τους, ακόμα χειρότερα προβλήματα επομένως. Πού να τα πουλήσουν αυτά. Άρα επομένως δεν υπάρχει ανιχνευσιμότητα, λένε οι, οι, οι οι κτηνοτρόφοι, κάποιο που είχε ας πούμε 500 και έχει τεράστια δαπάνη, αλλά τελικά είπε ότι προτιμούσε το παλιό σύστημα γιατί οι πλαστικέ ε, ετικέτε ήταν καλύτερε και ακόμη χειρότερα τα πράγματα στο σφαγείο γιατί εκεί πέρα έχουν ακόμη χειρότερο πρόβλημα για να δουν τι γίνεται. Ε, εκεί έχουν τα, τα νερά, έχουν θόρυβο τρομερό από τα εργαλεία του σφαγείου, οπότε το, το Bluetooth δεν μπορεί να διαβάσει την, την ετικέτα. Και, και η κατάσταση είναι ακόμα πιο μπερδεμένη όταν ε, προσπαθούν να πουλήσουν τα αρνιά τους, τα δικά τους που δεν έχουν ετικέτα, μαζί με αυτά που έχουν αγοράσει που έχουν ετικέτα, οπότε είναι μπερδεμένο. Άρα ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε πόσο μπερδεύτηκε η κατάσταση, γιατί ε, θα... Ε, δεν μπορούν να δουλέψουν. Οπότε παρακαλώ η Κομισιό να κάνει πίσω, γιατί νομίζω ότι τελικά οι καλύτεροι να διαχειριστούν την κατάσταση, νομίζω ότι είναι η ίδια κυβέρνηση της χώρας. George Lyon, σε la parola. George λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε και ο Τζιμ Νίκολσον, ο κύριο Λάιον, στα εξήγησε ότι δηλαδή έχουμε μια πάγια εκστρατεία κατά αυτού του μέτρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μαζί με τους συναδέλφους από τη Βόρεια Ιρλανδία δεν πετύχαμε και πάρα πολλά δεν μπορούσαμε να, να, να ανασχέσουμε την πορεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οπότε και ελπίζω ότι η, άρχισε η εφαρμογή και ίσως μπορεί να κάνει λίγο πίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να κάτσει να μελετήσει αναρωτώμενη μερικά πράγματα όπως το κατά πόσον αυτό το σύστημα και η δαπάνη του είναι ανάλογη με την ωφέλεια και με το σκοπό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει εδώ δυσαναλογία. Δεν, δεν ωφέλησε καθόλου πετυχαίνει αυτό το μέτρο το στόχο του. Εάν κάτσουμε και σκεφτούμε τι, τι, τι, τι feedback, τι εκθέσεις, τι, τι αναφορές έχουμε, ε, ε, νομίζω ότι η απάντηση είναι αρνητική. Ότι καταλήξαμε με, δύο διαφορετικά μητρώα όσον αφορά τις επιχειρήσεις, όσον αφορά το τι γίνεται στις ε, αγορές, ε, εκεί που πουλούνται τα αρνιά, ε, έχουμε πρόβλημα γιατί ο σκοπός ήταν ναι, να δυνατόν υπάρχει ανιγνευσιμότητα ε, με, με, με, με, ακρίβεια ιδίως σε περίπτωση κάποιας επιζωτίας όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται ούτε νομίζω ούτε έχω καταλάβει πως είναι το να πετύχει το μέτρο το στόχο του ε, γιατί νομίζω ότι όσον αφορά τα άλλα θέματα, το κατά πόσον αυτές οι έξτρα δαπάνες δικαιολογούνται, όσον αφορά ε, το, το, το, σκοπό και το όφελος πάλι εδώ έχουμε δυσαναλογία πάλι απάντηση είναι αρνητική άρα να αναρωτηθούμε το πιο βασικό είναι, υπάρχει σχέση ε, σωστή κόστους αποτελέσματος όχι επομένως θα πρέπει να δεσμευτεί η Επιτροπή ότι θα κάτσει και θα αναθεωρήσει την κατάσταση, να δει τι γίνεται με την εφαρμογή, έτσι να προσεγγίσει το θέμα. Να, να μην προχωράει στα τυφλά, γιατί τελευταία πενταετία εξαιτία αυτό έχει γίνει. Δεν κάθονται καν να ακούσουν τις προτάσεις των ε, εμπλεκομένων. Να γίνει επομένως μια ανοιχτόμυαλη διαδικασία και εξέταση για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα, να γίνει πιο αναλογικό, το, να υπάρχει καλή σχέση κόστος αποτελεσματικότητας, να πετύχει το στόχο του. Και αυτό πρέπει μια υπόσχεση της Κομισιόν ότι θα κάτσουν και θα μελετήσουν μια τέτοια διαδικασία ανθεώρησης. Τώρα το τελευταίο όσον αφορά κάποιες κυρώσεις και πρόστιμα πάρα πολύ στη Σκοτία είναι απελπισμένοι, ανησυχούν όσον αφορά τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται ή απειλούνται σε σχέση με διάφορες ε, παραβιάσεις για, για ε, υπέρβαση ορίων ε, σε σχέση με, με την cross compliance και βλέπουμε ότι είναι δύσκολο για αυτή τη τεχνολογία για να συμμορφωθεί κανείς και επομένω ε, είναι δυσβάχτατες αυτέ οι δαπάνε να πληθούν σε κάποιον ε, κτηνοτρόφο και περιμένω να μου πει σήμερα η Επιτροπή ότι κατανοεί ότι υπάρχει το πρόβλημα και ότι θέλει να δοθεί τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής μια ευελιξία όσον αφορά αυτές τις χρηματικές ποινές και τα πρόστιμα να γνωρίζει τη δυσκολία της υλοποίησης και αυτό γιατί υπάρχουν κάποια κουσούρια σε αυτό το σύστημα και υπάρχει δυσκολία εφαρμογής του. Αυτά ήθελα να σας πω και αυτέ αυτές τις δύο υποσχέσεις που σας είπα θα να ακούσω σήμερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι αυτό το σύστημα δεν είναι το πιο δόκιμο για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός. Παρακαλώ να περιορίσετε λίγο. Κυρία Ντότζ. Περιορίστε λίγο τι παρεμβάσει σα. Thank you, uh, Mr. President. I'm not sure that that uh, should be automatically directed at me, just as I Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι απευθύνεστε κατευθείαν σε μένα. Ευχαριστώ την Επιτροπή που ήρθε εδώ σήμερα διότι όπως πολλοί συνάδελφοι με ανησυχεί πάρα πολύ το θέμα αυτό διότι το καλοκαίρι παρακολούθησα διάφορες ε, εκθέσεις γεωργικές στη Βόρειο Ιρλανδία όπου είδαμε πολύ εμφανές το θέμα και ε, μεγάλη ανησυχία για αυτό το θέμα. Εξού και πιστεύω ότι περισσότερο περισσότεροι βοσκοί στους οποίους ε, μίλησα σκέφτονται να εγκαταλείψουν την, ε, ε, τον τομέα αυτό διότι όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν το φόβο των κυρώσεων από την πολλαπλή συμμόρφωση και δεν θέλουν να αναλάβουν αυτό τον κίνδυνο φοβούνται ότι θα υπάρξουν διάφορα πρόστιμα και έχουν έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια <coughs> και γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν έτσι και ανησυχούν πολύ με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα το οποίο δεν έχει συζητηθεί μέχρι στιγμής. Ότι δηλαδή εάν υπάρχουν πολύ περισσότεροι γεωργοί οι οποίοι εγκαταλείψουν τον τομέα αυτό τότε μπορεί να εγκαταλειφθεί και η γη και αυτό είναι πραγματικός κίνδυνος και πραγματικό πρόβλημα. Επίσης πολλοί γεωργοί έθεσαν θέμα ευημερία, πράγμα το οποίο αναφέρεται και εις πρόβλημα με ε, ε, ε, σκισμένα και μολυσμένα αυτιά των ζώων, τα προβλήματα που έχουν ήδη ήδη αναφερθεί επαναλαμβάνονται όσον αφορά την αξιοπιστία της αναγνώσεως και της διοικήσεως και της διαχειρήσεως που χρειάζεται ένα τέτοιο θέμα. Λοιπόν, όπως ο George Lyon ζητώ να υπάρξει μία αναθεώρηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί λογική και πρακτική λύση διότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα εις την καθυστέρηση ε, της ε, σημάνσεως μέχρι ότου το ζώο ετοιμάζεται να φύγει από την ε, εγκατάσταση για να ε, μην κοστι... Ε, επιβαρύνουμε το κόστος ιδίως για τους εξαγωγείς με την διεργασία αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνης έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επιτροπή. Θέλω να ε, προσθέσω μερικά σχόλια. Ε, δεν νομίζω ήταν σωστό ότι προχωρά η Επιτροπή στην ηλεκτρονική αναγνώριση τη στιγμή που η τεχνολογία δεν είναι εξασφαλισμένη. Θα ήθελα γραπτός να μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της πολλαπλής συμμόρφωσης, διότι είναι ένα πολύ οξύ θέμα για τους παραγωγούς και πρέπει ε, να αναγνωρίσουμε ότι οι γεωργοί ε, ε, ε, υφίστανται κυρώσεις για ατέλειες του συστήματος. Τώρα φαίνεται ότι στην Ιρλανδία έχουμε δύο συστήματα, ένα χειρονακτικό και ένα ηλεκτρονικό και αυτό θα οδηγήσει σε σύγχυση και αύξηση του κόστους για τους παραγωγούς προβάτων και πιστεύω ότι αν το σύστημα αποτύχει και υφίστανται οι κυρώσεις επίσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντές έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα σχόλια δείχνουν τι παράλογες διατάξεις πρέπει να εφαρμόσουμε. Γι' αυτό και έχω τέσσερις σύντομες ερωτήσεις στην Επιτροπή. Αν πρέπει να υπάρξει σήμηση, σήμαση εκατομμυρίων ζώων, ποιος θα υπεξεργαστεί τα, αποτελέσματα και τι κέρδος θα έχουμε. Τι θα γίνει αν το σύστημα δεν λειτουργεί. Εάν η, τρίτον, εάν η Ευρώπη καταφέρει να, να προβεί στην ηλεκτρονική αναγνώριση, τότε η ε, Επιτροπή θα απαγορεύσει την εισαγωγή ε, κρέατος από χώρες όπου δεν υπάρχει αυτή η ηλεκτρονική ανάγνωση και ε, τέταρτον με λίγο χιούμορ τα πρόβατα δεν ζουν σαν άδεια, άγρια ζώα εννοείται δηλαδή ότι και για τα άγρια ζώα θα προβούμε σε μια τέτοια ηλεκτρονική αναγνώριση. για να διευκρινίσω ότι δεν ανησυχούν μόνο οι Βρετανοί συνάδελφοι και εγώ έχω στη Γερμανία πολλά παράπονα από ε, καλλιεργητές και ε, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της θεωρίας και των καθημερινών προβλημάτων διότι οι εκτροφείς δέχονται εάν υπάρχουν ε, μικρές εκμεταλλεύσεις να, το, να συμμορφωθούν αλλά στα μεγάλα κοπάδια ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί και πρέπει να πούμε ότι οι βοσκοί ε, επίσης ε, προστατεύουν το περιβάλλον και δεν ε, πληρώνονται για το έργο αυτό το οποίο εκτελούν και το υψηλό κόστος εδώ δεν έχει σχέση με το κέρδος που αποκομίζουν από τα ζώα. Εάν λοιπόν ε, δεν ε, υπάρξει μια καλύτερη επίλυση των προβλημάτων δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ και δίνουμε το λόγο στην Επιτροπή τον κύριο Τομάντα που πρέπει να απαντήσει σε διάφορα θέματα και ελπίζω ότι θα απαντήσει σε όλους τους συναδέλφους. Θα προσπαθήσω να μιλήσω αγγλικά ώστε να μειωθούν οι παρανοήσεις. Καταρχήν όσον αφορά την αναλογικότητα. Πρέπει να επανέλθω στον λόγο ο οποίος οδήγησε στην υιοθέτηση ε, του κανονισμού 21 του 2004 ήταν μια κρίση που είχε οδηγήσει σε μεγάλες οικονομικές ζημιές, σε αυτοκτονίες στην Αγγλία και οδήγησε σε μια μετάδοση της ασθενείας από την Αγγλία στην Ιρλανδία και από εκεί μέσω Ολλανδία στην Ευρώπη διότι δεν μπορούσε κανείς να καταγράψει τις κινήσεις των εγωπροβάτων. Ε, ε, γυρίζω πίσω σε εκείνη την εποχή γιατί τότε ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια όλοι ζητούσαν ένα σύστημα σαφούς παρακολουθήσεως για να αποφύγουμε ε, το πρόβλημα του 2001 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και επανέρχομαι σε αυτό το γεγονός διότι διαφορετικά δεν καταλαβαίνόμαστε όταν μιλάμε. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ε, ε, εκλήθη να εφαρμόσει μέτρα, είναι ο θεματοφύλαξ των συνθήκων και ανέλαβε μέτρα με τη στήριξη του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εφαρμόσει αυτό το κανονισμό και πρέπει να πω ότι η τελευταία πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προέβλεπε την ε, ε, χρήση κάποιας ημερομηνία ή προθεσμίας για την ηλεκτρονική αναγνώριση. Είπε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας μετά ε, από την αξιολόγηση των προσόντων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απεφάσισε ε, στα πλαίσια που συζητάμε τώρα 1η Ιανουαρίου 2010 1η Ιανουαρίου 2011 πολλές φορές νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μία αμυντική στάση ενώ θέλει να είναι ε, χρήσιμη και να λύσει τα προβλήματα πρέπει όμως να εξασφαλίσει ότι ε, θα εφαρμόσουμε την νομοθεσία γιατί αυτό είναι και το καθήκον της στις περισσότερες χώρες δεν δεν έχουν ε, ε, σημειωθεί σοβαρά προβλήματα και αυτό είπα στην εισαγωγή ε, εάν δεν είχαμε προβλήματα ή στις μεταφράσεις. Αλλά μας έχουν αναφέρει διάφορα προβλήματα τα οποία φαίνονται να είναι εξαιρέσεις και όχι κανόνας. Κανείς δεν έχει μιλήσει μία ένα ποσοστό 20% αποτυχίας του συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ευχαρίστως θα δεχθεί την ε, πρόσκληση της κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου να επισκεφθεί τη χώρα ε, την επόμενη εβδομάδα και δεν νομίζω ότι θα μας πούν ότι δεν ξέρουν τι γίνεται στη χώρα τους. Όσον αφορά το πρόβλημα της ευημερίας μας ε, έχουν ε, αναφέρει προβλήματα στα νέα ζώα όταν υπάρχουν ε, σοβαρά σχισίματα και θα τα εξετάσουμε. Αλλά έχουμε δει ότι και για τα συνήθεια νότια υπάρχει τέτοιο πρόβλημα διότι υπάρχουν μύγες και άλλα ζωήφια που το καλοκαίρι μολύνουν τα πρόβα και γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα με όλα τα ενότια. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο θα καταγράφει όλες τις κινήσεις των εγωπροβάτων και θα μπορέσει να εντοπίσει την κίνηση του κάθε ζώου σύμφωνα με το, ε, την αρχή της ιχνηλασιμότητος που είναι ήδη ε, μέρος του κανονισμού του Συμβουλίου ε, και του Κοινοβουλίου υπαριθμών 178 για την ιχνηλασιμότητα στη διατροφική αλυσίδα. Επίσης αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι να αποφύγουμε με ασθένειες εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, να είναι ασφαλής η διακίνηση των ε, ζώντων ε, ζώων. Αυτό είναι ο στόχος του συστήματος. Όντως το σύστημα αυτό δεν απαιτεί από τις τρίτες χώρες να το εφαρμόσουν. Πρώτον, διότι βεβαίως δεν μπορούμε να υποχρώσουμε τις τρίτες χώρες να εφαρμόσουν την ε, νομοθεσία μας, ε, παρόλο που ε, εμείς αποφασίζουμε για τους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης όσον αφορά τα ζωντανά ζώα το ποσοστό εισαγωγών είναι αμεληταίο. Εάν δηλαδή δεν λάβουμε υπόψη την, ε, ε, την ε, Ελβετία που έχει τους ίδιους τους ε, ισότιμους κανόνες όπως εμείς και την Ορβηγία που έχει τους ίδιους κανόνες με μας. Ε, έχουμε ε, ελάχιστα ζώα τα οποία εισέρχονται ετησίως εκτός ε, από την Νορβηγία και την Ελβετία. Βέβαια όταν υπάρχει εισαγωγή κρέατος από εγωπρόβατα δεν έχουμε τους ίδιους κανόνες αλλά εμείς προσπαθούμε εδώ να εξασφαλίσουμε την ασφαλή διακίνηση των ζωντανών ζώων. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόζεται η νομοθεσία. Το Συμβούλιο και ε, το Κοινοβούλιο αποφάσισαν να υπάρξει μια ε, ατομική, ένα σύστημα ατομικής αναγνωρίσεως και ε, αυτό προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε χωρίς να δημιουργηθούν υπερβολικά προβλήματα. Ξέρουμε ότι το σύστημα είναι φιλόδοξο και ενδεχομένως στην αρχή της εφαρμογής σου θα προκαλέσει προβλήματα προσπαθούμε να τα περιορίσουμε, δεν θέλουμε οι κτηνοτρόφοι ε, στην μεταβατική φάση που δεν θα λειτουργεί σωστά το σύστημα να μην πληρώνουν οι κτηνοτρόφοι γι' αυτό, να μην πληρώνουν δηλαδή ε, κυρώσεις. Ε, θα δούμε και πώς θα εφαρμοστεί το σύστημα στην πρακτική και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, δόκτωρα Αλντομάτα. Τα προβλήματα είναι ακόμα πολλά, περίπλοκα, αλλά συμβάλαμε προσπαθώντας να κατανοήσουμε πού βρίσκονται τα πράγματα. Και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε, λοιπόν. Περνάμε στο επόμενο σημείο μας τώρα, στο 5. Α, όχι, ο George Λάιον θέλει να πανελθεί. Παρακαλώ, George. Ναι, θα ήθελα να ξεκαθαριστεί κάτι για αυτό το οποίο είπε στο τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν ανακοίνωση. Υπόσχονται ότι θα υπάρξει κάποιο πάγωμα επιβολής προστήμων. Έτσι κατάλαβα. Έτσι κατάλαβα, έτσι νόμιζα ότι άκουσα αυτό θα παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι έτσι όμως. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα δύο φορές στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά την επισήμανση των βοηδών. Έχουμε εκδώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την συμμόρφωση ή τις διατάξεις. Και εδώ πέρα υπάρχει μια σημαντική αρχή που ισχύει. Ότι όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα για τα οποία θεωρείται υπεύθυνο ο κτηνοτρόφος τότε αυτός δεν θεωρείται υπόλογος για το πρόστιμο. Παράδειγμα, Όπω γνωρίζετε όσον αφορά την επισήμανση των βοηδών θα πρέπει να υπάρχει διπλή ετικέτα στο αυτή. Ακριβώς γιατί ξέρουμε ότι ίσως χαθεί μια ετικέτα και άρα θα αρκέσει άλλη ούτως ώστε να ταυτοποιηθεί το ζώο. Επομένως υπάρχει υποχρέωση διπλής σήμανσης. Και γνωρίζουμε ότι ανάλογα με τις συνθήκες ε, της, εκμετάλλευση ότι μπορεί να χάσουν πολλά ζώα, τη μία ετικέτα και ίσως και τις δύο. Αυτό δεν είναι τόσο πιθανό, αλλά μπορεί να ισχύσει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, σε συνεργασία με τους αδέλφους Γενικής Διεθνής για τη Γεωργία, αποφασίσαμε ότι όταν αυτά γίνουν υπό συγκεκριμένες λογικές συνθήκες, που οδηγούν στην απόλυση ετικέτας, τότε δεν θα πρέπει να κληθεί να καταβάλει το πρόστιμο ο χνιοντρόφος. Όταν όμω μπει κάποιο σε μια εκμετάλλευση και 75% των ζώων έχουν μόνο μία ετικέτα και 20% καμία ετικέτα, ε, τότε υπάρχουν υποψίε ότι δεν εφαρμόζει την νομοθεσία ο κτηνοτρόφος. Φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου. Επομένως εμείς εδώ έχουμε εισαγάγει υπομορφή κατευθύνων γραμμών αυτή την αρχή. Επομένως, επειδή μέχρι σήμερα δεν είχαμε προβλήματα για, αυτή, για τη συμμόρφωση, την πολλαπλή συμμόρφωση, Μέχρι τώρα δεν είχαμε τίποτα δεσμενή συνέπειε. Τα συζητήσαμε με του συναδέλφου τη Γεωργία για το πώ αυτή η αρχή θα μπορέσει να ισχύσει σε, ένα διαφορετικό πλαίσιο, δηλαδή για τα σχετικά με την ηλεκτρονική και όχι συμβατική αναγνώριση. Επομένω, αυτό σα υποσχόμεθα. Θα το μελετήσουμε και θα σα πούμε, εάν είναι δυνατόν, τα τη αναγνώριση των βοηδών που εφαρμοστούν και εν προκειμένου. Πολύ καλά λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Από τώρα μπορούμε να περάσουμε, αν δεν δει άλλο το λόγο, στο επόμενο σημείο τη σημεία σα διάταξης. Σχετικά. Πολιτικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τι αναπτυσσόμενες χώρε προ ανάπτυξη τη πρόκληση τη επισητιστικής ασφάλεια. Θυμάστε, είχαμε ήδη συζητήσει για αυτό το θέμα μετά από την ανταλλαγή απόψεων τη τελευταία ε, συνεδρίαση. Το σχέδιο γνωμοδότηση του κυρίου Μάρκ Ταραμπέλα υπάρχει πλέον σε όλες τις ε, γλωσσικές εκδοχές. Θα δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στον κύριο Ταραμπέλα για να μας ενημερώσει και να σας θυμίσω ότι η υποβολή τροπολογιών ορίζεται για τις 14 Οκτωβρίου. 14 Οκτωβρίου στις 12 και όχι στις 25 Οκτωβρίου. Υπήρχε ένα λάθος στην προηγούμενη ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Μάρκετ Ταραμπέλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως θυμήσατε, είχαμε ήδη την ευκαιρία να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω πως ήταν στις 29 Σεπτεμβρίου όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό. Να σας πω εξ ότι Εάν τολμούσα να ξαναγράψω αυτή την έκθεση σήμερα θα την τροποποιούσα ήδη κάπως. Διότι καταρχήν ε, ξαναδιαβάζοντας την ανακοίνωση της Επιτροπής και είναι αλήθεια ότι η παράγραφος 1 της έκθεσής μου εκφράζει την χαρά της για την, για την Κομισιόν και για την πρότασή της. Ε, θα ήθελα να τη συγχαρώ γιατί η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει διάφορες ε, προβληματισμούς αλλά και προτάσεις ώστε να διορθωθούν ε, τα κακό σκήμενα όπως μέσω μιας καλύτερης συνεργασίας των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών που υπάρχουν ΦΑΟ, ΕΠΑΜ και ΦΙΝΤΕ. αλλά και επειδή δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Το θέμα της πείνας και της κακής διατροφής, ε, το λέμε εδώ και καιρό, δεν δλύνεται, αντίθετα επιδεινώνεται. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο ένα δις ανθρώπων, ακόμα και αν μιλάμε για 925 εκατομμύρια. Μπας περιπτώσει, εγώ πέρσι άκουσα για ένα δις ανθρώπων που υποφέρουν από σοβαρή κακή διατροφή. Ένα σωρό προγράμματα έχουν αναπτυχθεί, έχουν αποφασιστεί, ακόμα και G20 ασχολήθηκαν με το θέμα. Όλοι ασχολούνται με το θέμα. Η πολιτική αναπτυξιακή μα ε, ήταν ε, βέβαια μία από τι πιο αποτελεσματικέ στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει είμαστε από αυτού και το λέμε και το ξαναλέμε συχνά ότι είμαστε ανάμεσα στου μεγαλύτερου δωρητέ, αν προσθέσουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Ωστόσο παραμένει το πρόβλημα και ε, επιδεινώνεται. Έλεγα λοιπόν στην αρχή ότι αν χρειαζόταν να ξαναγράψω την έκθεσή μου, θα την έγραφα διαφορετικά σήμερα. Και άρα είμαι ανοιχτό στη συζήτηση με τους συναδέλφους και ειδικά τους όδης εισηγητές, αλλά και όλους τους υπολείπους γιατί όπως είπατε Πρόεδρε είναι η 14η Οκτωβρίου το μεσημέρι η προθεσμία για την υποβολή των τροπιών βέβαια πολλές τροπολογίες θα λάβουμε γιατί με βάση τις συζητήσεις που κάνουμε Ήδη είδαμε ότι υπήρχαν αντιδράσεις που μάλιστα ήταν θετικές τόσο απέναντι στην έκθεσή μου όσο και απέναντι στην ανακοίνωση της Επιτροπής που θέλω και πάλι να αντιχαιρετήσω διότι προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι προσπάθησα όλα αυτά να τα συνοψίσω σε καμιά δεκαριά σημεία, δεν χρειάζεται να τα θυμίσω όλα γιατί ήδη τα έχουμε συζητήσει αλλά νομίζω πως έπρεπε να θυμίσουμε ότι η γεωργική ανάπτυξη θα πρέπει να βασίζεται στο δικαίωμα να μπορεί κανείς να τρέφεται από τρόφιμα, με τρόφιμα και ότι η τροφική ε, κυριαρχία των κρατών είναι εγγυημένη από την Ένωση. Να θυμίσουμε επίσης ότι η πιο στερημένοι λαοί ε, θα πρέπει να δημιουργήσουν μια γεωργία, γεωργία ε, επιβίωσης, ε, δηλαδή δεν πρέπει να παράγει ζωοτροφές, γιατί εδώ αναφέρω ένα παράδειγμα, γιατί εδώ δεν κάνουμε διπλωματία, κάνουμε πολιτική. Όταν μαθαίνουμε, ας πούμε, ότι η Νιγηρία είναι μια χώρα με ένα μεγάλο πρόβλημα, πρόγραμμα για την ε, ανάπτυξη της καλλιέργειας φίνικα ε, για παραγωγή ελαίων για βιοκαύσιμα. Είχαμε ήδη την Ιδονησία και τη Μαλαισία, ενώ το 29% των παιδιών που υποφέρουν από κακή διατροφή σε αυτή τη χώρα και 12 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ιγυρία φέρνουν από πίνε και αυτοί βάζουν palm oil tree, δηλαδή φίνικες για παραγωγή ελαίων μόνο, για καύσιμα, για βιοκαύσιμα. Ίσως λοιπόν αυτό πρέπει να τα συζητήσουμε με τις ενισχύσεις αναπτυξιακές που ε, τους δίνουμε, να λαμβάνουμε υπόψη τις αποφάσεις που ε, παίρνουν αυτές οι χώρες, αφού ο βασικός στόχος είναι να χορτάσουν οι πληθυσμοί. Ε, και σίγουρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τις περιφερειακές ε, εμπορικές συμφωνίες ε, για να ευνοηθούν οι τοπικές παραγωγές και να υπάρξουν ανταλλαγέ ανάμεσα σε χώρες που είναι πλέον ασματικές σε ορισμένες παραγωγές και ελληματικές σε κάποιες άλλες ανά περιφέρειες του κόσμου, ώστε να μην μετακινούνται μακριά τα προϊόντα στις τοπικές αγορές, να διοχετεύονται και στις περιφερειακές και να λειτουργούν αυτά παραπληρωματικά, να συμπληρώνουν οι γείτονες μεταξύ τους τις παραγωγές τους, αν αυτό είναι εφικτό να διασφαλιστεί η, σε παγκόσμιο επίπεδο οι πιο βιο, οι, να διασφαλιστούν οι πιο βιώσιμες και λιγότερο ενεργοβόρες μέθοδοι παραγωγής Ίσως επίσης να μην είχαμε μια διαφορετική εκτίμηση όσον αφορά την αγγλική μετάφραση. Να επιμείνω για το γεγονός ότι η μη διατροφική χρήση των υλικών προϊόντων και όπως ας πούμε τα βιοκαύσιμα θα πρέπει εδώ να προσέχουμε και να βάλουμε όρια γιατί σε, στο εγγύς μέλλον Μπορεί να βασιστούμε στις ε, πετρελαιοπαραγωγικές εταιρείες που μας λένε ότι εξαντλούνται οι πόροι, εξαντλούνται τα πετρελαϊκά κοιτάσματα. Φυσικά, αν υπήρχε και θα υπάρξει στο μέλλον σίγουρα υπάρξει αύξηση των τιμών των στερεών καυσίμων, είναι σαφές ότι θα πρέπει να, υπάρξουν, να θέσουμε ασφαλιστικές δικλείδες και να μην στραφούμε σε μια γεωργική παραγωγή υποκατάστατων που θα βλάψει την ε, παραγωγή τροφίμων που μας απασχολεί σήμερα. Τώρα, πρόσβαση στη γη. Ξέρουμε ότι οι ορισμένες χώρες της Αφρικής αλλά και η Ασία, η Νότια Ασία υποφέρει από κακή διατροφή. Αλλά σε εστιαστούμε στην Αφρική, γιατί από τα 830 εκατομμύρια που ζουν εκεί, τα, τα, 240 υποφέρουν από κακή διατροφή. διατροφή. Ε, ε, είναι επίσης μια ήπειρος που είναι υπό ε, όπου γίνεται εκ νέου απεικιοποίηση. η Κίνα αυτή τη στιγμή απικίζει την Αφρική, την ξανά απικίζει σίγουρα τουλάχιστον κάποιες χώρες. Όπως σας είπα δεν μιλάμε εδώ διπλωματικά, μιλάμε για πολιτική και παράγει για εξαγωγή εκεί στην Αφρική και όχι για να στηρίξει τις τοπικές ανάγκες. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε με κατάρτιση για να κινήσουμε τους νέους, να μπορέσουν να, να επενδύσουν στην παραγωγή την γεωργική και έτσι να διατηρηθεί ένας πληθυσμό στις ε, γεωργικές περιοχές, περιοχέ της υπαίθρου, να αποφευθεί η αστιφιλία και φυσικά να επιμείνουμε στην ενίσχυση της έρευνα ε, από δημόσια κεφάλαια και τη διάδοση της νόησης στον τομέα της βιώσιμης ε, γεωργίας αλλά και την έρευνα γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην εξέλιξη των εισοδημάτων όπως την γνωρίζουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη από ό,τι σε, άλλες, σε άλλα μέρη του κόσμου που είναι αλήθεια πως η έρευνα θα μπορούσε να βοηθήσει στην πλήρωση ορισμένων ελλημάτων της παραγωγής. Όλοι γνωρίζουμε ότι το 2050 θα χρειαζόμαστε μια γεωργική παραγωγή διπλάσια Πράγμα το οποίο δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει όσον αφορά τις τροφικές συνήθειες και την εξέλιξή του στι αναδυόμενε χώρε. Ακόμα και αν πρόκειται μόνο για γνωμοδότηση, ίσω θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε για να στείλουμε ένα ε, έντονο μήνυμα, ένα ισχυρό μήνυμα, ώστε οι συνάδελφοι να προσ... αν το είχα ξαναγράψει μάλλον θα δεχόμουν το... και κάποια κείμενα της Κομισιόν και θα τα είχα βάλει εδώ ώστε να υπάρξουμε, να έχουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν θα ακρηγορήσω άλλο. Ευχαριστούμε Μάρκ. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό και σε ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σου. Και τώρα ξεκινάμε την συζήτηση με τον Λουίς Καπούλα Σάντος που ζήτησε τον λόγο. Έχουμε διάφορους που ζήτησαν τον λόγο και εδώ θα προσπαθήσουμε να οργανωθούμε σωστά. Παρακαλώ Λουίς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν να συγχαρώ τον συνάδελφο Μάρκ για την ποιότητα της εργασίας του που είναι άλλωστε συνηθισμένη. Ε, αυτή που περιμένουμε από εκείνον. Ωστόσο υπάρχει κάποιο έλλειμμα και που νομίζω υπάρχει και στην ανακοίνωση του Ισκομισιόν και είναι το πρόβλημα της διαχείρισης, της διακυβέρνησης, γιατί το κεντρικό πρόβλημα από την άποψη το, της διατροφής για πολλές χώρες που υποφέρουν από αυτό το πρόβλημα είναι πρόβλημα διακυβέρνησης. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να ε, πάντα αναλυστικά αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όταν εμείς έχουμε μια άσχημη, κακή, μάλλον βεβαρημένη συνείδηση όσον αφορά την απεικιοκρατία, και να τους πούμε πώς θα πρέπει να διαχειριστούν τα πράγματα εκεί, αλλά είναι ένα κεντρικό πρόβλημα. Και ο Μάρκο το, το ανέφερε πριν από λίγες μέρες, είδα ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει ότι μία από τις χώρες στο κέρας της Αφρικής τα παιδιά πάνε σχολείο στα κινέζικα. Η πρώτη τους ε, επαφή με το σχολείο και με τη γραπτή γλώσσα είναι τα κινέζικα. Μα είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να μας αφήσει διάφορους. Δεν θέλουμε να να υποκαταστήσουμε μια νέα μορφή απεικιοποίηση. αλλά εν πάση περιπτώσει όσο και σωστή και αν είναι η ανακοίνωση τη Κομισιόν και όσο και είναι σωστή η έκθεση του συναδέλφου Μάρκ Ταραμπέλα, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το κεντρικό θέμα που είναι το θέμα τη διακυβέρνηση. και θα να δούμε αν θα έχουμε και αρκετή φαντασία για να προτείνουμε κάποιες τροπολογίες που να καλύψουν αυτό το έλλειμμα, την έλλειψη αυτή. Πολύ δύσκολο βέβαια να είναι κανείς καλύτερος από τον Μάρκ. Σας ευχαριστώ, Λουίς. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρά το πρόβλημα. Ο Στεφάν Λεφόν έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις σχετικά με ε, τις ε, καλλιέργειες επιβίωσης. Ε, ήθελα να ε, ξέρω εάν αυτό ε, αντιτίθεται ή στις εξαγωγικές καλλιέργειες, διότι καταρχήν ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, τις τοπικές τις τοπικές αγορές η Αφρική δεν πρέπει ε, να ε, καταδικαστεί να έχει μόνο μία καλλιέργεια επιβίωσης ε, πρέπει να παράγουμε ε, ε, για την εσωτερική αγορά και μετά για, την εξαγωγή, για τις εξαγωγές. Επίσης θα πρέπει να ξαναεπενδύσουμε στη γεωργία για να την αναπτύξουμε διότι ε, πιστεύαμε πολύ καιρό ότι το θέματα αυτά θα λυνόντουσαν με τις με ε, τις ε, ανταλλαγές, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και θυμάστε ότι στο στην προηγούμενη θητεία μας είχαμε δυσκολία να πείσουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε για να μπορέσουν τα κράτη να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους. Άρα και η Ευρώπη πρέπει να θεωρήσει ότι η Γεωργία είναι μία προτεραιότητά της. Πολύ καλά. η Ραντς Ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι το 2050 θα έχουμε 70% επιπλέον ανάγκες διατροφικές. Άρα το θέμα αυτό μας απασχολεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο εξαρτώμαστε από το εξωτερικό, όλο και περισσότερο έχουμε ένα σύστημα ανταλλαγής υλικών ε, ε, και διατροφικών ε, ειδών με προϊόντα από τις τρίτες χώρες. Οπότε το να διαθέσει κανείς ένα δισεκατομμύριο δολάρια για τις υποανάπτυξη χώρες είναι αξιέπαινο αλλά πρέπει να δούμε αν μπορούμε να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις περιφέρειες περιφέρειες διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι Ευρωπαίοι υποφέρουν από τις διακυμάνσεις των, ε, και την αστάθεια των τιμών. Οπότε ε, όταν αγοράζουμε ε, τεράστιες εκτάσεις στις ανάπτυξη χώρες. Το συζητούσαμε ε, όταν μιλούσαμε για την Αφρική και τις εξαγορές των Κινέζων. Ε, θα πρέπει ίσως και εμείς να ανησυχήσουμε και ε, να αντιμετωπίσουμε την ε, αντίφαση που υπάρχει μεταξύ των ανησυχιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλά για το μέλλον για επαρκή διατροφή τη στιγμή ε, που δεν ενισχύει την παραγωγή εντός της Ευρώπης. Πρέπει να αναθεωρήσουμε την ΚΑΠ και ε, να ε, ασχοληθούμε ε, με το μέλλον στα πλαίσια του εγγράφου που θα παρουσιαστεί στις 17 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ. Μάρτιν Όσλινγκ. Καταρχήν συμφωνώ με την έκθεση του Μάρκ Ταραμπέλα. Πιστεύω ότι αναφέρονται όλα τα σημαντικά στοιχεία και υπάρχει ένα θέμα ακόμη που πρέπει να εξετάσουμε, να ε, κηρύξουμε ότι είμαστε κατά κάθε πολιτικής dumping των τιμών διότι έτσι καταστρέφονται πολλοί γεωργοί στις τρίτες χώρες οι οποίοι συνέρχονται με τα μεγάλες δυσκολίες ή δεν συνέρχονται ποτέ. Ε, λοιπόν, ε, με τις ε, ενισχύσεις πιέζει κανείς ορισμένες αγορές και οι εντόπιοι μικροί γεωργοί δεν έχουν πλέον καμιά δυνατότητα. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή έδειξε ότι ουσιαστικά η διατροφή εξασφαλίζεται από τους μικρούς γεωργούς και πρέπει να στηριχθεί η προσπάθειά τους. Γι' αυτό ε, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μία περικοπή σημαντική των πιστώσεων και δεν μπορούμε πλέον να επενδύσουμε στον τομέα αυτό, ε, δεν είναι καθόλου σωστό. Ε, είναι λοιπόν ένα θέμα που πρέπει να παραμείνει στη μερίσια διάταξη και δεν πρέπει να μας απασχολεί μόνο η Κίνα που μας ανησυχεί, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε και εμείς τις μεγάλες άλλες γεωργικές επιχειρήσεις μας ε, που προωθούν τα βιοκαύσιμα τα οποία δεν αγοράζονται καν σε ορισμένες χώρες. Πρέπει λοιπόν να ε, ε, ε, δεν είναι δυνατόν να επηρεάζει κανείς τις αγορές κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι καλύτερες εκτάσεις στις τρίτες χώρες να αναφέρονται για την καλλιέργεια βιοκαυσίμων. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα αλλά υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να έχουν στις περιφερειακές αγορές φθηνά τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα. Η κυρία Γέγκλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Μάρκ για την εισαγωγή και για όλους, και όλους τους προλαλήσαντες για τα προβλήματα τα οποία έχουν περιγράψει και τα οποία διαβλέπω. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στην πολιτική κατάσταση γιατί χωρίς σταθερή πολιτική κατάσταση στις διάφορες χώρες την οποία πρέπει να πετύσουμε θα μιλάμε χρόνια και τίποτα δεν θα βελτιωθεί, θα γίνεται απλώς πιο δύσκολο. Επίσης πιστεύω ότι είναι σωστό ότι χρειαζόμαστε μικρότερες δομές και θα πρέπει να επιτρέψουμε ε, να υπάρξουν και μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Θα πρέπει να μπορούν οι γεωργοί αυτοί να κερδίσουν χρήματα, να ε, θρέψουν την οικογένειά τους, αλλά να μπορούν να επενδύσουν επίσης. Βλέπω ότι υπάρχει ένα σύνολο και η διατύπωση ότι προωθούμε με την ε, τοπική ε, γεωργία είναι πολύ ε, εύστοχη θα ήθελα επίσης να πω ότι οι κράτη-μέλη και Ευρωπαϊκή Ένωση ή και άλλοι που χρηματοδοτούν ορισμένες περιοχές θα πρέπει να ε, ε, τους ζητήσουμε να σκέφτονται περισσότερο τη γεωργία από ό,τι το έχουν πράξει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα κενό το οποίο πρέπει να καλύψουμε στον τομέα αυτό. Και θέλω τελικά να πω ότι την περασμένη Πέμπτη ψηφίσαμε στην Ολομέλεια μία έκθεση σχετικά με την βιοπικιλότητα στις υποανάπτυξη χώρες όπου με μεγάλη ε, πλειοψηφία δεχθήκαμε μία τροπολογία η οποία ε, ε, είναι τελεί, ίδια και απαράλλαχτη ε, με την ε, ε, πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και επιρρύπτει ευθύνε για τα προβλήματα των υποανάπτυξη χωρών. Καλό λοιπόν θα ήταν και στο σημείο αυτό η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική να διατυπωθεί κατά τέτοιον τρόπο όπως είναι αρμόζων και όχι όπως ε, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία ε, σε αυτή την τροπολογία. Μας έκανε μεγάλο κακό ε, αυτό το οποίο κάναμε στην τροπολογία αυτή και νομίζω ότι και αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί περαιτέρω και σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Κάτι το οποίο τόνισα στην έκθεση στην τελευταία θητεία του Κοινοβουλίου για το ότι η κάπαλα και η ασφάλεια στα τρόφιμα ήταν το γεγονός ότι οι δαπάνες στην Γεωργία αλλά και η αναπτυξιακή βοήθεια είναι όλο και λιγότερο δαπανώνται στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπως είπε και ο συνάδελφος Λαφόλ. Πολύ σημαντική παρατήρηση για το θέμα της διακυβέρνησης. Πιστεύω πως η πολιτική κατάσταση είναι πολύ σημαντική. Δείτε τη Ζιμπάμπουε που υπήρχε πραγματικά ανθίζουσα γεωργία που έτρεφε όχι μόνο το λαό της Ζιμπάμπουε αλλά και άλλες χώρες και μέσω του πολι... λόγω του πολιτικού συστήματος κατέρευσαν τα πάντα. Πώς... Και τι μπορεί να κάνει η Ένωση να ενθαρρύνει αν η χώρα είναι ασταθής. Είναι πρόβλημα αυτό και πρέπει να το εξετάσουμε. Και οι ίδιε οι Αφρικανικέ χώρε πρέπει να θέσουν ω προτεραιότητα την ανάπτυξη τη γεωργία. Στηρίζω την παρατήρηση τη κυρία Γέγλε για την κλίμακα των ε, αγροκτημάτων. Εμένα, για μένα το θέμα αυτό δεν είναι πρόβλημα. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα διάφορα είδη <coughs> γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι να δώσουμε μια πολιτική βάση όπου οι αφρικανικές χώρες θα μπορέσουν να αναπτύξουν την γεωργία όσο γίνεται καλύτερα για τις ίδιες. Και αυτό σημαίνει σταθερή παραγωγή και σταθερές τιμές για τους παραγωγούς. Η Αφρική χρειάζεται μια κοινή γεωργική πολιτική. Γιατί λειτουργήσε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γεωργία ωστόσο θα πρέπει να, είναι ε, προτεραιότητα και για τις ε, ίδιες τις χώρες της Αφρικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Άρκεν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραμπέλα για την έκθεσή του. Ένα-δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω ακόμα. Μιλήσαμε για την οργάνωση και συμφωνώ με τον Χόσλινγκ ότι ο μόνος κόσμος που δεν πρέπει να κατονομάζουμε μόνο τους Κινέζους γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν μπλεχτεί στην απεικιοκρατία Πρόκειται για ένα παιχνίδι ε, ε, ισχύω και ε, επιρροής. Ε, θα πρέπει να δούμε και τη δύναμη, την ισχύ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πως αυτές και πολλές από αυτές κάνουν το ίδιο ακριβώς όπως και οι Κινέζοι στις ε, τρίτες χώρες και πολλοί από τους παραγωγούς εκεί βρίσκονται σε πολύ πιο αδύναμη θέση από τη γεωργία της Ένωσης. Αυτό είναι κάτι δεν πρέπει δεν να το ξεχνάμε και να το γνωρούμε. Μιλήσαμε κάπως για τη βοήθεια φαντάζομαι ότι είναι κάπως πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά κάποιος πρόσφατα πήγε στην Αϊτή να προσπαθήσει να βοηθήσει κάποιους από τους ε, πτυνοτρόφους ε, και παραγωγούς ε, αυγών και όταν αυτός ο άνθρωπος ήρθε πίσω είχε τελείως απογοητευτεί με το τι συμβαίνει, γιατί το σχόλιο του ήταν ότι ακόμα κι αν οι βοήθειες, η βοήθεια και οι υπηρεσίε βοήθειας εκεί είχαν καλές προθέσεις, δεν ήξεραν τίποτα για την κτηνοτροφία. Είναι πολύ σημαντικό αν είναι δυνατόν, να ευθυγραμμίζεται η βοήθεια με πραγματική εμπειρογνωμοσύνη, ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, να μην είναι μόνο να πούμε ότι θα κάνουμε κάτι, αλλά να διασφαλίσουμε και ότι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά. Τώρα, κάποιοι μίλησαν για την πολιτική κατάσταση. Και εντάξει, Μας είπε η Επιτροπή ότι δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η ανιχνευσιμότητα που μπορούμε να, μπορούμε να επιβάλλουμε στην Ένωση περιμένουμε να εφαρμοστεί και αλλού. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό, είναι αλήθεια, αλλά ε, το ίδιο ισχύει και για, τις, ε, για αυτή την περίπτωση. Και Μειώμενη στήριξη για τη γεωργία στην Ένωση. Αν δούμε τις ανάγκες για μια πλήρη παραγωγή στα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να πούμε δύο λόγια για το, σχέση, το, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασφάλιση της ασφάλειας κιόλα. Τε, ωραία, τελευταίος ομιλητής, τελευταία ομιλήτρια μάλλον, ε, ομιλητής ο κύριος Νταντέ. Και εμείς είχαμε μια παρόμοια, ένα παρόμοιο πρόβλημα με την έκθεση για την ΚΑΠ. Ξέρετε η έκθεση του συναδέλφου Λάιν που έλεγε ότι πρέπει να διατηρηθούν τα κονδύλια της ΚΑΠ. Και στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου, μετά από την πρωτοβουλία τη Επιτροπή ε, ανάπτυξη, ψηφίσαμε μια έκθεση που λέει τελείω τα αντίθετα. Καλό θα ήταν να κάνουμε μια έκθεση, λοιπόν, μια συνάντηση εργασία μαζί με την Επιτροπή ανάπτυξη για να τα αποψαφινίσουμε, γιατί πολλοί κόσμος παραμένει, πιστεύει σε κλισέ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και αυτή την παρέμβαση του Μισελ Νταντέν. Συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να κάνουμε μια δουλειά συντονισμού. Γιατί θα πρέπει αυτά όλα να συνδεθούν με το θέμα της τροφικής ασφάλειας, της επάρκειας ε, της διατροφικής. Και εμείς που συντάσσουμε τους κανόνες της μελλοντική γεωρικής πολιτικής ε, μετά το 2013, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι δίπλα από το θέμα της ποιότητας είναι και το θέμα της ποσότητας. Ε, πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο για να τα βάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε όλοι να καταλάβουν τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Επιτροπή, τον κύριο Όλτοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον κύριο Τεραμπέλα για την στήριξη στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Να σας πω ότι αυτή η ανακοίνωση αφορά την ασφάλεια τη διατροφική και η ώρα που χρησιμοποιούμε δεν είναι συμπτωματική και θα ήθελα να κάνω μια αποσαφήνιση γιατί στη συζήτηση εδώ χρησιμοποιήθηκε η, ο όρος τροφική κυριαρχία που είναι κάπως διαφορετικός και από ό,τι γνωρίζω πρόκειται για ορολογία που δεν έχει υποστηριχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφάλεια διατροφική είναι ο όρος που χρησιμοποιείται. Food security. Επίσης, η ανακοίνωση μιλάει για τις, ε, τα, τις εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας, όχι για, τη, για τα, τις εκμεταλλεύσεις επιβίωσης. Ε, θέλουμε να λυθεί το θέμα της πείνας. Η πείνα είναι κυρίαρχη στα συστήματα μικρό, όπου, όπου επικρατούν μάλλον οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Και γι' αυτό και στόχος της δημόσιας στήριξης θα πρέπει να είναι αυτός, αυτή η κλίμακα. Αυτό δεν σημαίνει ότι στον τομέα στον κόσμο μάλλον της ε, γεωργίας ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν υπάρχει χώρος για άλλου είδους άλλες κλίμακες, ε, όχι. Αλλά εμείς αυτό προτείνουμε όσον αφορά τη βοήθεια. Δύο, Δύο άλλα σημεία που θέλω να σας αναφέρω πρώτα πρώτα όσον αφορά το ότι κατά κάποιο τρόπο χάθηκε στη συζήτηση η σχέση μεταξύ του τι συμβαίνει από πλευρά γεωργία στην Ευρώπη και στον Αναψόνο από την μεριά. Εγώ θεωρώ ότι θα έχει εμβαθύνει περισσότερο από αυτού η Επιτροπή σας. Δεύτερη παρατηρήση αφορά την γεωργία και την Πίνα διότι η ανακοίνωση αναγνωρίζει ότι ακόμα και αν υπάρχει υπάρχει τροφίμων σε μια χώρα το θέμα της πείνας δεν είναι αυτονόητο ότι λύνεται άρα κανείς θα πρέπει να πάει πέρα από το θέμα της γεωργίας και των καλύτερων επιδόσεων της γεωργικής παραγωγής γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι που εφαρμόζονται η και περισσότερο στο τρίτο κόσμο που θεωρούνται παρέμβαση κοινωνικού δικτύου σε Ινδία, σε Αιθιοπία. Έχουμε αυτό το δίκτυ ασφαλείας και δεν χρειάζεται επομένω να παρέμβει κανείς μέσω της γεωργίας για να περιστύλει το πρόβλημα της πείνας και σας ευχαριστώ. Πολύ καλά λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Μάρκ Ταραμπέλα για τη δουλειά του και τώρα ε, θα δευτερολογήσεις για να κλείσει η συζήτηση είμαι πάρα πολύ σύντομος και πριν σας είπα ότι ότι αν το ξανά έκανα το ίδιο σήμερα, το ξανά έκανα διαφορετικά για να μπορέσω να περιλάβω στην έκθεση αυτά τα οποία ελέγχθησαν πρώτα-πρώτα ο, ο, ο που είπε ότι βεβαίως και υπάρχει πρόβλημα σε πολλές χώρες όσον αφορά τις επιλογές που έγιναν οπότε δεν είναι δυνατόν απομονωμένα να, να ενεργήσουμε για το πρόβλημα ή στην Γεωργία μόνο και όπως έλεγα στην αρχή είναι δυνατόν εδώ να, να πούμε πολλά αλλά αν θέλουμε να είναι το μήνυμα δυναμικό δεν θα πρέπει να απομονωθούμε μόνο στα της γεωργίας αλλά ούτε μπορούμε να ξεχάσουμε επομένω ε, το, το, το, το, τη γενικότερη συγκυρία γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και ε, έχουμε επίσης την Αρμόδια Επιτροπή της Ουσίας, την Επιτροπή Ανάπτυξης, οπότε θα πρέπει να τονιστεί και πάλι το ότι θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερε επενδύσει στα γεωργικά προγράμματα μέσω τη πολιτική ανάπτυξη. Δεν θα μακρηγορήσω, αλλά όπω σα προείπα, είμαι πρόθυμο να ακούσω πάσα πρόταση και επίσης πρόκειται τους ε, σκιώδη συζητά κάθε πολιτική ομάδας ε, να τους συμβουλευτώ και ξέρετε ότι μέχρι τις 14 Οκτωβρίου το μεσημέρι μπορείτε να κατεβάσετε κάποιες προτάσεις, θα τα πούμε και ενδεχομένως μπορούμε και να εκμετρευτούμε και το διάστημα της Ολομελίας στο Στασβού την επόμενη εβδομάδα, ούτως ώστε να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχεδόν εισηγητών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, τους ξέρουμε Πολύ ωραία λέει πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. τελειώσαμε αυτό το σημείο και πάμε τώρα στο σημείο 6 τη ημερησία διατάξεω που αφορά την εμπορία υλικών ε, αγενού πολλαπλασιασμού τη ε, Αμπέλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είπε ότι πρόκειται να στείλει την κωδικοποίηση οδηγία του 68 του 93 και διαπιστώθηκαν ότι υπάρχουν κάποια σημεία τη ουσία που θα πρέπει να αλλάξουν. Οπότε είπε ότι θα αλλάξει την κωδικοποίηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα κάνει ένα καινούριο κείμενο. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν άλλαξε τις, διατυπώσεις, τις διατάξεις σχετικές με την επιτροπολογία και βέβαια τώρα έχουμε ευρύτερε αρμοδιότητε με δυνάμει τη ειδική τη Λισαβόνα. Πρώτο θα το ο κύριο ε, Ταμπάτζη και κατόπιν η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ουσιαστικά το είπατε και εσείς και φαντάζομαι ότι τώρα η νομική επιτροπή ε, θα ε, ασχοληθεί με αυτή τη συζήτηση. Ε, για μας όμως πρόκειται πάλι για ένα θέμα νομικό και εφόσον δεν είμαστε νομικοί δεν μας χαροποιεί. Πρόκειται περί αυτού. Έχουμε ένα τραπέζι το οποίο παράγει ένας ξυλουργός με τέσσερα πόδια και κάθε πόδι έχει διαφορετικό μήκος και το τραπέζι αυτό παρήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε γιατί δεν είναι σταθερό. Άρα ο Μαραγκός, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή πρέπει να αποφασίσει εάν θα το επιδιορθώσει για να κόψει τα πόδια όλα στο ίδιο ύψος ή ε, εμείς θα ζητήσουμε ε, από τα κράτη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρουν πίσω το τραπέζι αυτό και να το επιδιορθώσουν. Δεν θέλω να επεκταθώ στην παρομοίωση αυτή, αλλά ε, θα πρέπει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιληφθεί ότι δεν έχει ενσωματώσει τη συνθήκη της Λισαβόνας και ε, δεν βασίζει τις αρμοδιότητές της στη συνθήκη της Λισαβόνας αλλά σε άλλες έννοιες και σε άλλες συνθήκες διότι εδώ βλέπουμε στην την επιτροπολογία που δεν υπάρχει πλέον υπάρχουν τα, οι εντεταλμένες νομικές πράξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αντιληφθεί ότι θα ήταν σκοπιμότερο να αποσύρει αυτή την αναμόρφωση του κτηρίου ή στη συνέχεια να αποφασίσει η Επιτροπή Γεωργίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή μάλλον ε, η το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξουν ορισμένα σημεία του κειμένου που δεν συνάδουν με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό είναι το πρόβλημα αγαπητοί κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ή θα αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να αποσύρει αυτή την ε, ε, νέα ε, έκδοση για να την συμμορφώσει στη συνθήκη της Λισαβόνας ή διαφορετικά θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να βρει τη λύση. Ωραία. Δίνω λοιπόν τον ε, λόγο στον ε, Δοκτώρ Τσιμάη. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν ορισμένα νομικά ζητήματα τα οποία ανέκυψαν από την τελευταία παρέμβαση. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να σας κουράσω στην Επιτροπή σας πόσο λίπες με τεχνικά θέματα να σας κουράσουν με αυτά τα νομικά. Καθαρά νομικά είναι. Απλώς με δύο λόγια να αναφερθώ στο ότι έχουν ακουστεί διαφορετικές απόψεις από το καθαρισμικό οργάνο σε σχέση με το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις ισχύουσες διατάξεις επιτροπολογίας. Το συμπέρασμα μας είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε καινούργια νομοθετήματα επί τη βάση αυτής της νέας ε, διαδικασίας, όμως θα μπορούμε τώρα να αναφερθούμε στις παλιότερες διατάξεις για την Επιτροπολογία. Για αυτές έχουμε κάποιες διαφορετικές απόψεις ε, το του Κοινοβουλίου, διότι θεωρείται ότι οι εκείνες διατάξεις δεν είναι δυνατόν να χρησιμεύσουν για νέα νομοθετήματα. Και Συμβούλιο και Επιτροπή πρεσβεύουν ότι αντίθετα είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να επικαλούμε αυτές τις παλαιότερες διατάξεις. Και έτσι να έχουμε νέες ομοθετικές πράξεις. Αυτά έως ότου προκύψει ένας νέος κανονισμός όσον αφορά τις εφαρμοστικές αρμοδιότητες. Όμως, όπως προείπα, θα προτιμούσα να είμαι σύντομος και να μην μακρηγορούμε όσον αφορά αυτές τις νομικές λεπτομέρειες. Θα προτιμούσα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε κάποια πιο πρακτικά θέματα. Από τη μία πλευρά τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει μια διαδικασία μελέτης για νομοθεσία τέτοιου είδους. Και αυτή η διαδικασία μελέτης και περίσκεψης ενδεχομένως καταλήξει σε κάποιες πρωτοβουλίες μεταρρυθμιστικές κατά το εγγύς μέλλον, ας πούμε ένα-δύο χρόνια. Α, του χρόνου, του χρόνου. Ναι, σωστά. Ευχαριστώ με διορθώνετε. Και υπάρχει επομένω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης μελετά το τι θα κάνει με αυτές τις διαδικασίες τη Επιτροπολογία οι οποίε περιέχονται στις ισχύουσε νομοθετικέ πράξει. Ε, ε. Και μιλούμε τώρα για τις ε, οριζόντιες μοναδικές ε, πράξεις. Για όλους αυτούς τους λόγους, όσον αφορά την συζητούμενη πρόταση, εμείς θα προτείναμε να ανασταλεί η νομοπαρασκευαστική διαδικασία εν αναμονή ενδεχομένων άλλων πρωτοβολιών οι οποίες ίσως αναλυφθούν. Ο Φερρυπίν ευρύτερη αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το τι θα γίνει με την επιτροπολογία η οποία θα ισχύει για το εν λόγω νομοθέτημα. Bene. Non so se, ε, tutto chiaro. Μάλιστα. Καταλάβατε όλα. Ο Ταμπάτζη. Ταμπάτζη θες να ξαναπάρεις το λόγο. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν ξανά το λόγο. Όχι. Εσύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέλω να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι αυτή είναι μια πολύ σοφή απόφαση δηλαδή εσείς θα κόψετε και θα ισιώσετε τα πόδια του τραπεζιού δεν έχει σχέση με αυτό το συγκεκριμένο θέμα αλλά στο σημείο αυτό είναι αρμόδια μόνο η Επιτροπή Γεωργία μόνο εμείς μπορούμε να δεχθούμε ή να απορρίψουμε αυτή τη διαδικασία αν πρόκειται για ένα νομικό θέμα. Ευχαριστώ. Eh, Μάλιστα. Αφού δεν υπάρχουν άλλε πατρίσει, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ταβάζη και να πάμε στο τελευταίο σημείο. Αυτό που προσθέσαμε απόψε και θα δώσω αμέσω το λόγο στην κυρία Μαγκίνε και μετά στον κύριο Λαβία που θέλουν να μα ε, μιλήσουν για το πρόβλημα του προπολογισμού. Μαγκίνες, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξέρω την αργά, αλλά θα είμαι σύντομη είναι ένα θέμα σε σχέση με μια συγκεκριμένη γραμμή του προπολογισμού. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Και βασικά είναι τα χρήματα που περιμένει η Κομισιόν να επιστρέψουν τα κρατημέλη λόγω αντασταλιών στον γεωργικό προϋπολογισμό. 72 εκατομμύρια περιμένει η Κομισιόν. Αλλά το Συμβούλιο υπολόγισε 492 εκατομμύρια. Κατά την άποψή μου, μέσω δημιουργικής λογιστικής βρήκαν 422 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια παραπάνω από την Κομισιόν. Εμείς στηρίξαμε τα στοιχεία της Κομισιόν με τη βάση της εμπειρίας των προηγούμενων ετών. Το πρόβλημα είναι πως τώρα στο προπολογισμό, στην Επιτροπή Προπολογισμού απορρίφθηκε η δική μας τροπολογία με μικρή πλειοψηφία και η Επιτροπή υποστηρίζει το νούμερο του Συμβουλίου, 492 εκατομμύρια. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται να επανυποβάλουμε τις τροπολογίες για την Ολομέλεια, διότι θα έχουμε πρόβλημα το 2011 αν παραμένει αυτός ο αριθμός. Και θα πρέπει να βρούμε ε, εξοικονομήσει από στον προπολογισμό του 2011, αν μείνει αυτό το νούμερο. Γι' αυτό και είναι επίγον να αξιολογήσουμε και τη γνώμη των υπολείπων και να, δούμε, να το σκεφτούμε και ίσως δώστε τα σχόλιά σας για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Πρέπει οπωσδήποτε να λύσουμε το πρόβλημα. Τζοβάνι. Πιστεύω ότι αυτή η πανυποβολή είναι απαραίτητη, γιατί με την νέα διαδικασία της συνθήκης της Λισαβόνας μπορεί να είναι η Κομισιόν η οποία επανυποβάλλει, η Επιτροπή μάλλον που επανυποβάλλει μια τροπολογία που έχει απορριφθεί, γιατί η Επιτροπή μας είναι που την είχε υποβάλει. Αλλά πάντως πιστεύω πως το Συμβούλιο, επειδή δεν θέλει να κάνει περικοπές σε συγκεκριμένες γραμμές του προπολογισμού, αποφάσισε να μειώσει συνολικά το γεωργικό προπολογισμό κατά 420 εκατομμύρια ευρώ. Ε, Κατά τη διάρκεια της χρήσης βέβαια κατά τη δυνατότητα να πάει να βρει από πού θα αφαιρέσει τα ποσά αυτά. Αυτή είναι μια στρατηγική την οποία έχει, ε, ήδη έχει προσπαθήσει να επιβάλλει το Συμβούλιο στο παρελθόν και πιστεύω ότι η Επιτροπή Γεωργίας και οι διάφορες πολιτικές ομάδες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επανεπιβάλλουν τροπολογία και να την υπερψηφίσουν. Για να σας δώσω μια ιδέα είναι ε, ότι αν δεν αποκατασταθεί αυτό το σχέδιο του προπολογισμού θα καταλήξουμε στο, η πρόταση που προκύπτει από το Κοινοβούλιο, που προέρχεται μάλλον από το Κοινοβούλιο για το νέο γεωργικό προπολογισμό, να είναι ένας προπολογισμό ε, που έχει περικοπεί σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, παρά τις προσθήκες που έχουμε κάνει, κατά τόσα εκατομμύρια ευρώ. Εμείς ως Κοινοβούλιο περιοτείνουμε πιο περιορισμένο προπολογισμό σε σχέση με αυτόν που στην πράξη είχε υποβάλει η Κομισιόν. Γι' αυτό και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να αποκαταστήσει, η Επιτροπή μας δηλαδή, θα πρέπει να αποκαταστήσει αυτή την τροπολογία και να ζητήσει από όλε τι πολιτικέ ομάδε ε, στην Ολομέλεια να τη στηρίξουν. Γιατί νομίζω πω υπήρξε και κάποια σύγχυση ανάμεσα στι ε, πολιτικέ ομάδε στον ε, Επιτροπή Προπολογισμού. Κάποιο κατάλογο ψηφοφορία δεν ήταν σύμφωνο με την κοινή λογική και αίσθημα των συναδέλφων. Ευχαριστώ, Τζοβάνι. Ο Τζορτζ Λάιον ζήτησε το λόγο. Εγώ, εξ ονόματο τη ομάδα μου, εγώ λοιπόν ε, υποστηρίζω την ε, εκ νέου υποβολή τη τροπολογία και ε, θα φροντίσω ώστε ο κατάλογος ψηφοφορία της ομάδας μου να είναι σωστός και θα τους συμβουλεύσω να το υπερψηφίσουν. Και από τους σοσιαλιστές από ό,τι κατάλαβα υπήρχε κάποιο προβληματάκι. Ναι, να δώσουμε γρήγορα το λόγο στον Λουίς Καπούλας Σάντος. Εμείς εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας είχαμε αποφασίσει για μια θέση και αυτή διατηρούμε. Όπως γνωρίζετε πολλές φορές δεν είναι δυνατόν μέσα στην ίδια ομάδα την πολιτική να είμαστε όλοι σύμφωνοι και στην Επιτροπή Γεωργίας και στην Επιτροπή του Προϋπολογισμού. Στη... σοσιαλιστές εδώ, πάντως στην Επιτροπή Γεωργίας, θα διατηρήσει τη θέση που κράτησε και στην προηγούμενη ψηφοφορία και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προσπαθήσει να πείσει την πλειοψηφία των συναδέλφων να μας στηρίξουν. Μάλιστα. Και εγώ το προσυπογράφω αυτό. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις συμφωνούμε από ό,τι κατάλαβα όλοι να το επανυποβάλλουμε όλοι στο όνομα της Επιτροπής. Δεν χρειάζονται οι 40 υπογραφές και θα το ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Άρα λοιπόν δέσμευση όλων να περάσουμε αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ Μάριον, ευχαριστώ Τζοβάνι. Τέλος της συνεδρίασης. Very